Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Με μεγάλη χαρά σα καλωσορίζω στη συνεδρίαση τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού που συνεχίζεται από χθε. Έχουμε φέτο την παρουσίαση των ετήσιων εκθέσεων του Ελεκτικού Συνεδρίου και χαιρετίζω την παρουσία του Προέδρου του ελεκτικού συνεδρίου, καθώς και ορισμένων μελών του ελεκτικού συνεδρίου. Η ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου είναι για μας ως Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού πέραν της διαδικασίας ε, απαλλαγής το σημαντικότερο γεγονός του έτους. Εμείς βασιζόμαστε στα πορίσματα του Ελεκτικού συνεδρίου γιατί μας δίνει πραγματικά τη δυνατότητα να δούμε καλύτερα πώς λειτουργούν οι διοικητικές δομές στην ε, Κομισιόν, στις, στους αποκεντρωμένους φορείς και επίσης και η σχέση όλων αυτών των οργανισμών και των φορέων με τα κράτη-μέλη. Έχουμε επίσης παρόντα τον Επίτροπο κ. Σεμέτα, ο οποίος είναι ο συνομιλητής μας για τα θέματα ελέγχου του προπολογισμού από την πλευρά της Κομισιόν. Προτείνω λοιπόν να περάσουμε κατευθείαν στην έκθεσή σας, κύριε <clears throat> Καλτέιρα, και στη συνέχεια μπορούμε να έχουμε την υποβολή ερωτήσεων. Έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, Επίτροπε, αξιότιμα μέλη, αγαπητέ εισηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε την έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή του προπολογισμού και το, για το Ταμείο Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή τη Ανάπτυξη, οι πολίτε τη Ευρώπη έχουν το δικαίωμα να ξέρουν πώ δαπανούνται τα χρήματά του και κατά πόσο χρησιμοποιούνται σωστά και κατά πόσο τους δίνει ε, αξία τη στιγμή όπου υπάρχει η περικοπή στα δημοσιονομικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χειρίζεται πρωτίστω του πόρου Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δίνει πληροφορίε για τα λογιστικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση yeah. και πώ χρησιμοποιούνται οι πόροι. Και πόσο κανονικά γίνονται οι οικονομικέ διαδικασίε και ποια είναι τα αποτελέσματα. Το ελεκτικό συνέδριο που αξιολογεί ανεξάρτητα τα τρία αυτά στοιχεία της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως της οικονομικής διαχείρισης σύμφωνα με τη συνθήκη και τα επαγγελματικά πρότυπα για τον έλεγχο και τις βέλτιστες πρακτικές. Παρουσιάζει το ελεκτικό συνέδριο το αποτέλεσμα του εξολογήσεως της εφαρμογής του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην ετήσια έκθεσή του, ούτως ώστε να βοηθήσει το Κοινοβούλιο ε, στην διαδικασία της απαλλαγής το κεφάλαιο 1 της ετήσιας έκθεσής μας παρέχει ε, τη δήλωση εξοπιστίας όσον αφορά την, ε, το βάσιμο των λογιστικών και την κανονικότητα των διαφόρων ε, οικονομικών συναλλαγών. Τα κεφάλαια 2 μέχρι 9 αξιολογούν τα έσοδα και τους βασικούς τόμους τις βασικές δαπάνες και το κεφάλαιο 10 ε, είναι αφορά τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, λοιπόν, ποια είναι η εξολόγηση του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενώσης του 2012. Η γενική εικόνα μοιάζει κατά πολύ με την εικόνα της εκθέσεως της Περσινής. Υπάρχουν όμως κάποια ιδιαίτερα σημεία στην ετήσια έκθεση που θα ήθελα να τα τονίσω και να επιστήσω την προσοχή των μελών της Επιτροπής. Και αυτά τα σημεία σχετίζονται με τέσσερα βασικά θέματα. Πρώτα απ' όλα την ομιμότητα και την τακτικότητα των πληρωμών. Δεύτερον, οικονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις. Τρίτον, η πίεση επί των δημοσιονομικών της Ευρωπαϊκής και τέλος την ανάγκη να δημιουργηθεί μια, ένας πολιτισμός επιδόσεων κατά την ε, περίοδο του επομένου δημοσιονομικού πλαισίου. Θα ξεκινήσω με την γενική εικόνα. Τα λογιστικά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι αξιόπιστα όπως ήταν από το 2007 τα έσοδα και ανάληψη υποχρεώσεων και είναι όλα τακτικά και κανονικά από ηλικής πλευράς. Οι πληρωμές όμως εξακολουθούν οι υλικά να επηρεάζονται από την όλη κατάσταση. Όσον αφορά την επίδειξη αποτελεσμάτων από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ακόμα σε θέση να δώσει επαρχή σχετικά και αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά τα επιτέγματα των ευρωπαϊκών πολιτικών και με τρόπο που να είναι καλός για τη διαδικασία της απαλλαγής. Η άποψη του ελεκτικού συνέδριου στην φαινομιμότητα και την τακτικό χαρακτήρα των πληρωμών έχει παραμείνει η ίδια εν γέννη διότι δείχνει και ποια είναι υποβόσκουσα πραγματικότητα που δεν άλλαξε σημαντικά. Το ελεκτικό συνέδριο εκδίδει αντίθετη γνώμη σύμφωνα με τα στοιχεία από τους ελέγχους και από την αξιολόγηση των διαφόρων συστημάτων ελέγχου και από ε, δειγματοληπτικά στοιχεία των συναλλαγών. Εξετάσαμε τα ελεγχτικά συστήματα και είδαμε ότι είναι μόνο αποτελεσματικά, μερικά αποτελεσματικά όσον αφορά την νομιμότητα και το ευτικό χαρακτήρα των πληρωμών όταν οι δαπάνες πραγματοποιούνται της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Βάσει της δοκιμής κάποιων δειγμάτων συναλλαγών φρονεί το Ελεκτικό Συνέδριο ότι το επίπεδο ασφαλμάτων για τις πληρωμές δαπανών και στα λογιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 4,8% το περιθώριο ασφαλμάτων. Το Ελεκτικό Συνέδριο είναι 95% σίγουρο ότι το ποσοστό ασφαλμάτων στις πληρωμές κοίται μεταξύ 3 και 6%. Αυτά τα σφάλματα δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένους τομείς του προπολογισμού, όλες οι ομάδες πολιτικών που καλύπτουν σε επιχειρηματικές δαπάνες επηρεάζονται υλικά από το σφάλμα και οι διοικητικές δαπάνες είναι ο μόνος τομέας όπου δεν έχουμε πραγματικό επίπεδο σφαλμάτων, υλικό επίπεδο σφαλμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εκθέσεις της επιβεβαιώνει τη γενική εικόνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται ότι τα σφάλματα πραγματοποιούνται σε όλα τα σημεία του προπολογισμού και έτσι έχει κατάσταση. 14 γενικές διευθύνσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν επιφυλάξει όσον αφορά τι αιτήσει εκθέσει δραστηριοτήτων, όσον αφορά την ομιμότητα και τακτικό χαρακτήρα των δαπάνων. Και οι συνοπτικές εκθέσεις δείχνουν ότι το επίπεδο του σφάλματος είναι μεταξύ 1,9 και 2,6% των συνολικών πληρωμών. Ένα στοιχείο που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι πιθανότατα αποτελεί υποτίμηση όπως βλέπετε από το κεφάλαιο 1, η γενική εκτίμηση του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά το πιθανό επίπεδο ασφαλμάτων αυξήθηκε από 3,9 που ήταν το 2011 στα 4,8 το 2012. Το ελεκτικό συνέδριο εκτιμά ότι το πιθανό επίπεδο ασφαλμάτων για τη γεωργία, περιφερειακή πολιτική, απανάπτυξη πέθρου, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις δείχνει αύξηση εν συγκρίση με το 2011 ανάψη πέθρου εξακολουθεί να έχει τα περισσότερα σφάλματα στον αφορά τις δαπάνες. Περίπου 7,9% είναι το ποσοστό των σφαλμάτων και μετά έχουμε την περιφερειακή πολιτική με 6,8%. Υπάρχουν και αυξήσει στα σφάλματα που εκτιμούνται για την έρευνα και άλλες εσωτερικές πολιτικές και για τις εξωτερικές σχέσεις και βοήθεια και διεύρυνση. Σε αυτές τις περιστάσεις ένα τμήμα της αύξησης μπορεί να αποδοθεί σε δύο μεθοδολογικές βελτιώσεις που εισήγαγε για το ελεκτικό συνέδριο για τον έλεγχο του 2012. Τα δείγματα συναλλαγών του ελεκτικού συνεδρίου στους δύο αυτούς τομείς δεν συμπεριλαμβάνουν τις μεταβατικέ πληρωμές που έγιναν κατά διάρκεια του έτους. Με άλλα λόγια, οι διάμεσες πληρωμές, τελικές πληρωμές και προκαταβολές του έτους. Αυτές οι αλλαγές σύμφωνα με τη γραμμή των αναλογιστικών κανόνων δίνουν μια καλύτερη εικόνα της πραγματικότητας όσον αφορά τα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η δεύτερη μεθοδολογική βελτίωση σχετίζεται με την εντόπιση των σοβαρής, σοβαρών σφαλμάτων εφαρμογή κανόνων περί κρατικών προμηθειών. Το 2012 οι θεσμικοί φορεί τη Ευρωπαϊκής Ενώσεως αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών και άλλοι διεθνείς φορείς. Αυτές οι αλλαγές βελτιώνουν τη συγκρισιμότητα μεταξύ των διαφόρων ομάδων πολιτικών και βελτιώνουν τη συγκρισιμότητα με την πάροδο του χρόνου. Όλα αυτά μαζί προσθέτουν 0,3% στη Γενική Εκτίμηση του λεκτικού Συνεδρίου όσον αφορά το πιθανό επίπεδο σφαλμάτων για το 2012 εν συγκρίση με το 2011. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η ετήσια έκθεση του Εκτικού Συνεδρίου του 2012 συμπεριλαμβάνει πολλά παραδείγματα όσον αφορά τα σφάλματα που ευρέθησαν και γίνεται και σημαντική ανάλυση από αυτών. Όλα αυτά μαζί δίνουν κάποια εικόνα για το πού προκύπτουν τα σφάλματα και πώς επηρεάζουν την κατάσταση. Επιτρέψτε μου να δώσω μερικά παραδείγματα όσον αφορά την ανάλυση που παρέχουμε στην έκθεση. Καταρχάς, πάνω από δύο τρίτα των εκτιμωμένων ποσοστών σφαλμάτων αφορούν τη μη επιλεξιμότητα των αξιώσεων για πληρωμές και σοβαρά λάθη στον αφορά την εφαρμογή των κανόνων περί δημοσίων προμηθειών. Δεύτερον, μεγαλύτερη συνεισφορά στα ασφάλματα αφορά τους τομείς όπου εκεί θα παρούν τα περισσότερα χρήματα, δηλαδή περιφερειακή πολιτική, γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, απασχόληση και κοινωνικά θέματα. Τρίτον, το ελεκτικό συνέδριο δοκίμασε διάφορε συναλλαγέ και εκεί είδαμε ότι το ποσοστό των συναλλαγών που επηρεάζονται από τα σφάλματα είναι πολύ υψηλό σε αυτούς τους τομείς πολιτικών. Από 35% μέχρι 63% το επίπεδο σφαλμάτων. Και τέταρτον, η δοκιμή συναλλαγών του ελεκτικού συνεδρίου δείχνει ότι πάνω από τα μισά σφάλματα που βρήκε το ελεκτικό συνέδριο και στα πλαίσια της κοινή διαχείρισης θα μπορούσαν να είχαν διορθωθεί μέσω εθνικών δράσεων από τις εθνικές αρχές πριν υποβάλουν αξιώσεις για επιστροφές χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα πορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου δεν διατείνονται ότι περιορίζονται σφάλματα σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Στην πραγματικότητα, εξολόγηση των εποπτικών συστημάτων έδειξε ότι υπάρχουν αδυναμίες σε ευρύ φάσμα διαφόρων φορέων εθνικών και περιφερειακών. Ούτε τα σφάλματα περιορίζονται στις δαπάνες και μόνο που αποτελεί τμήμα τη κοινή διαχείριση με τα κάτι μελη Υπολογίζει το ελεκτικό συνέδριο ότι το εκτιμόμενο ποσοστό σφάλματο όσον αφορά την κοινή διαχείριση των δαπανών ήταν 5,3% εν συγκρίση με το 4,3% σε όλε τι άλλε μορφέ ε, των δαπανών στα πλαίσια συνεργασία. Τα σφάλματα που βρίσκεται στο ελεκτικό συνέδριο έχουν σημασία ότι προσωπεύουν περιπτώσει όπου οι πόροι τη Ευρωπαϊκή Ενώση χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ότι ο τρόπο δεν συνάδουν με τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που είναι νομοθέτες και δημοσιονομική αρχή. Και έχουν σημασία τα σφάλματα, δείχνουν ότι αυτά τα χρήματα δεν έπρεπε να πληρωθούν, να καταβληθούν. Καμιά φορά αληθεύει ότι είναι δυνατόν αυτά τα χρήματα να ανακτηθούν. Και εδώ έρχομαι στο θέμα των οικονομικών διορθώσεων και των ανακτήσεων. Το ελεκτικό συνέδριο ε, αφιερώνει πολλές παραγράφους στην τέτοια έκθεσή του για το 2012 σε αυτό το θέμα. Ε, είναι περίπλοκο το ζήτημα και το Ελεκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσεγγίζουν από διαφορετικέ αλλά συμπληρωματικέ ε, πορείε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να προστατεύσει τον προπολογισμό από τι συνέπειε των μετασταλιών. Το Ελεκτικό Συνέδριο είναι υποχρεωμένο να αναφέρει κατά πόσο οι συναλλαγέ είναι νόμιμε και τακτικέ. Το 2012 η ετήσια, στην ετήσια έκθεση διερευνάται από το Ελεκτικό Συνέδριο πώς γίνονται οικονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις στα κατημέλη. Τι σημασία έχουν αυτές ανακτήσεις στους τελικούς δικαιούχους και σχετικά με αφορά τις δηλώσεις, δηλώσεις Οι διορθώσεις εξαρτώνται από τους εφαρμόσιμους κανονισμούς. Παραδείγματο χάρη για τη γεωργία, τις περισσότερες οικονομικές διορθώσεις δεν οδηγούν τα κάτι μελη να ανακτήσουν πληρωμές από τους δικαιούχους. Ενώ για τη συνοχή οι περισσότερες διορθώσεις είναι διορθώσεις που δεν οδηγούν σε λεπτομερή ε, διόρθωση σε επίπεδα προγραμμάτων. Έτσι, ε, οι περισσότερες οικονομικές διορθώσεις εμπίπτουν σε εθνικά πλαίσια και το τονίζει αυτό το εκτικό συνέδριο. Η τρίσια έκθεση απευθύνεται και προς τις εθνικές αρχές και τα εθνικά κοινοβούλια. Πρόεδρε, μέλη, προσπαθώντας να βελτιώσουμε την οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν μπορούμε να γνώσουμε την αυξανόμενη πίεση όσον αφορά τα δημοσιονομικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το ελεκτικό συνέδριο τονίζει ότι αυξάνεται η πίεση επί του προβλησμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την πραγματοποίηση των πληρωμών στην έκθεση του 2012. Όπω γνωρίζετε, το 2012 η Επιτροπή ήδη αντιμετώπιζε δυσχέρειε όσον αφορά την κάλυψη όλων των ετοιμάτων πληρωμή. Η πίεση επί των πληρωμών αντανακλάται επίση στην αύξηση του ποσού των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων. Στο τέλος του 2012 αυτές αντιστοιχούσαν σε περισσότερα από δύο έτη των συνολικών πληρωμών της Ευρωπαϊκή Ενώσεω που καταχωρίζονται ως δαπάνες. επίση, η Επιτροπή θα χρειαστεί να χρηματοδοτήσει πληρωμέ προκειμένου να καλύψει υποχρεώσει στον ισολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Στο τέλο του οικονομικού έτου 2012, οι εκκρεμεί αναλήψει υποχρεώσεων και υποχρεώσει που έχριζαν χρηματοδότηση ανερχόταν από κοινού σε 313 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Κατά τη γνώμη του συνεδρίου, η Επιτροπή πρέπει να σχεδιάζει τι μελλοντικέ απαιτήσει για ταμιακέ ροέ, καταρτίζοντα και δημοσιεύοντα μια μεγάλη κλίμακα πρόγνωση για τι ταμιακέ ροέ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, δεν είναι πάντοτε υπεύθυνοι οι ηθοποίοι για την ποιότητα των επιδόσεών τους σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόβλημα εντοπίζεται στο σενάριο που τους δόθηκε. Τα ισχύοντα νομικά πλαίσια για τις δαπάνες δεν ενθαρρύνουν επαρκώς τη βελτίωση της ποιότητας των δαπανών. Η περίοδος του νέου δημοσιονομικού πλαισίου παρέχει την ευκαιρία να αλλάξει η κατάσταση αυτή. Το συνέδριο συμφωνεί με την Επιτροπή ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας μιας νοοτροπίας προσανατολισμένης στις επιδόσεις. Αυτό σημαίνει ότι μετοπιστούν οι αδυναμίες που διαπιστώνει το συνέδριο στο ισχύον σύστημα διαχείρισης και της εκθέσεων, παραδείγματος χάρη σε τρει βασικού τομεί. Τα προγράμματα δαπανών δεν χρησιμοποιούν με συνέπεια στόχους ε, ούτε κατάλληλου δείκτε. Τα δεδομένα σχετικά με τι επιδόσει είναι λοιπού ποιότητα και υπερβολικά συχνά τα έργα που χρηματοδοτούνται με δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω δεν είναι βιώσιμα. Είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά αν η επόμενη γενιά προγραμμάτων δαπανών πρόκειται να παρέχει και να είναι φανερό ότι παρέχει προ τη θέμενη αξία στην Ευρώπη και του πολίτε τη. Το συνέδριο συνιστά εστίαση στι επιδόσει για την ερχόμενη περίοδο προγραμματισμού. Αυτό απαιτεί τον καθορισμό σαφών στόχων συναφών δικτών και προσδοκόμενων αποτελεσμάτων. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρειαστεί να συνεργαστούν για τη βελτίωση των επιδόσεων και της λογοδοσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα επόμενα έτη. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, μέσω των ετησίων εκθέσεών του, συνέβαλαν και θα συμβάλλουν και θα συνεχίσουν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτυχία του, του συλλογικού αυτού εγχειρήματο. Προσβλέπουμε στο να ξεκολουθήσουμε, να διαδραματίζουμε το ρόλο μα από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των λοιπόν θεσμικών οργάνων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καλντέιρα για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλά σημαντικά σημεία και πρωτού δώσω τώρα το λόγο στον αρμόδιο επίτροπο τον κύριο Σεμέτα για να λάβει και αυτός θέση από την οπτική γωνία της Κομισιόν. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω εμάς με Y κύριε Καλντέιρα για την πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή μας σε ό,τι αφορά την ετήσια έκθεση. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια μεγάλη ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ πληρωμών και υποχρεώσεων. Αυτά τα λεγόμενα ραλ, τα τα λικιντέ είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τα μάλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί κατεπηγόντως και σε ό,τι αφορά την αποτελεσματόστροφη διαχείριση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει τονίσει και ο ίδιος ο εισηγητής και πολλοί άλλοι στην Επιτροπή μας. Το θέμα λοιπόν του εκτιμόμενου ποσοστού σφαλμάτων είναι ένα ποσοστό το οποίο φαίνεται ότι έχει αυξηθεί, ενώ εμείς νομίζαμε ότι τα πράγματα βελτιώνονται. Και δεν έχουμε καταφέρει να μειώσουμε <clears throat> αυτό το ποσοστό σφαλμάτων. Αυτό φυσικά δεν είναι κάτι το οποίο οφείλεται μοναχά στην ευθύνη των φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εμπίπτει και στην αρμοδιότητα και την ευθύνη των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θέλαμε λοιπόν να έχουμε την άποψη του κυρίου Σεμέτα, ο οποίος ενδεχομένως μπορεί να μας ε, διαφωτίσει σε ορισμένα από τα ερωτήματα που έχει θέσει ο πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου. Κύριε Επίτροπε, σας δίνω το λόγο λοιπόν. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ισηγητά, Πρόεδρε Καλντέρα, αξιότιμα μέλη της ε, Επιτροπής ελέγχου προπολογισμών και του ελεγκτικού συνεδρίου. Η δημοσίευση της ετησία εκθέσεως του ελεγκτικού συνεδρίου είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη καμπή της διαδικασίας απαλλαγής του προπολογισμού. Είμαστε ευγνώμες για αυτό το τιτάνιο έργο το οποίο ακόμα μια φορά επιτελέσατε και επίσης ε, θεωρούμε πάρα πολύ θετικά τα συμπεράσματά σας και τις ε, συστάσεις σας. Οπότε και δεν μπορούμε παρά να χαιρετήσουμε το ότι το συμπέρασμα σας είναι ότι ε, δεν έχουμε ε, λάθη ανακριβείς ε, εγγραφές και ότι το ποσοστό όσον αφορά τα σφάλματα για τα διοικητικά, για τα έσοδα είναι κάτω από το όριο σημαντικό του το 2%. Επίσης, οι υποχρεώσεις σε κάθε ε, δαπάνη ε, επίσης πήραν το πράσινο φως και γι' αυτό έχουμε την ε, ανάντη προετοιμασία των προγραμμάτων, των έργων, των χορηγήσεων και των συμβάσεων που χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία. Επίσης, φέτος έχουμε μάλλον την αύξηση του ποσοστού σφάλματος για τις πληρωμές. Ε, και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια καινούργια νοοτροπία όσον αφορά τις επιδόσεις μας και γι' αυτό κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις που θα συζητηθούν στο Στασβούργο όσον αφορά το MFF. Και επίσης θεωρούμε ότι το ποστό σφάλματος για τις πληρωμές και την εκαθάριση της προχρηματοδότηση του 2012 στο 4,4% για πληρωμέ εκείνη του έτου σε σχέση με το 3,9% του 2011. Και όπως και εσείς είπατε, το 1 τρίτον τη αυξήσεω σχετίζεται με την καινούργια μεθοδολογία ε, τη δειγματοληψίας όσον αφορά τι άμεσε πληρωμές και το απομένον 0,6% ε, θα αντισταθμιστεί από κάποιο είδους ε, πάγιες διορθώ, πάγιες ή κατά αποκοπή διορθώσεις που τις επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν ε, τα κράτη-μέλη υποβάλουν τις ε, αξιώσεις τους και που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Ελληνικό Συνέδριο και ε, διαχρονικά έχετε θεωρήσει ότι, ότι αυτά είναι οι πηγές και οι αιτίες των ασφαλμάτων και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, πώς αυτά θα τα συγκρατήσουμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο και όσον αφορά τα προγράμματα που έχει στο κρατημέλη, το Ελληνικό Συνέδριο επιβεβαιώνει ότι οι παραβάσεις των εθνικών ε, διατάξεων είναι η αιτία για ένα σημαντικό ποσοστό όσον αφορά ε, το συνολικό ποσό του φάρμαντος και γι' αυτό και εμείς έχουμε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την ε, απλούστευση, τόσο να αντικαταστήσουμε τα εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητα που είναι περίπλοκα και έτσι θα έχουμε ε, άλλου είδους ε, επιλογές όσον αφορά τις δαπάνες γιατί τη σήμερα ημέρα έχουμε τα απλουστευμένες επιλογές δαπανού 20% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του 2012 δεν διαπιστώσατε εσείς τίποτε σφάλματα σε σχέση με αυτού του είδους τις, ε, τις κινήσεις ε, και όσον αφορά τις υπόλοιπες δράσεις του Κοινωνικού Ταμείου, η συχνότητα του σφάλματος ήταν 40%. Και όσον αφορά τον τομέα της έρευνας, είχαμε πει ότι θα συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα Horizon 2020 και ο χρυσός κανόνα θα είναι ένα πρόγραμμα και μία χρηματοδότηση. Έτσι να είναι η χρηματοδότηση ευκολότερη και γι' αυτό και έχουμε καταποκοπή ε, διαχείριση των εμέσων δαπανών το οποίο έτσι ε, θεσπίστηκε. Και επίσης ε, θεωρούμε ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί σε σχέση 2011 και έχουμε ακόμα υψηλά ποσοστά ασφαλμάτων για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα έχουμε αυτού του είδους τους κανόνες διαχείρισης που είναι περίπλοκοι και κάποιες χώρες όπως η και Ιταλία έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες ε, αν συγκριθούν με άλλα κράτη-μέλη που έχουν λίγα λειτουργικά προγράμματα και ενδιάμεσους οργανισμούς και φορείς. Επίσης είδαμε ότι ο έλεγχος των ε, δαπανών ε, δεν γίνεται με αποδοτικό τρόπο και έτσι έχουμε ακόμα περισσότερα λάθη. Επίσης έχουμε τυπολατρία αντί για ουσιαστικό έλεγχο. Δεν έχουμε έλεγχο των κανόνων που διέπουν τις δημοσίες συμβάσεις και διαγωνισμούς και επίσης υπάρχει πίεση πιστοποίηση των δαπανών για να μην έχουμε ε, κάποιο είδους διακοπής χορήγησης των κονδυλίων και επίσης υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τις δυνατότητες της διοίκησης και τους πόρους αυτής. Επίσης, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει για να προσθέσουμε τους κανόνες σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις δηλώσεις των δαπανών ε, να δούμε τι συγκεκριμένα θα κάνουμε εμεί ω Κομισιόν. Έχουμε μια αυστηρή πολιτική όσον αφορά τι διακοπές και τι αναστολές και είπαμε ότι όταν δούμε ότι υπάρχει επανάληψη των ίδιων αδυναμιών, σταματάμε τι πληρωμέ. Το 2011 είχαμε 91 διακοπέ και 2,6 ευρώ, το 2012 είχαμε 116 διακοπέ και έφτανε αυτό στα 5 δις ευρώ περίπου. Οι δεπληρωμές ξεκινούν και πάλι μόνο αφού γίνει μια ερευνητική πραγμάτων επιτροπή και, ε, και γίνει και οικονομικό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μόνο αν οι ε, η αρμόδια για τον οικονομικό έλεγχο αρχή έχει πιστοποιήσει ότι τα προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί ε, επαρκώ. Κατά δεύτερο λόγο, το 2013 εμεί κάναμε θεματικού οικονομικού ελέγχου, τόσο να μπορέσουμε να εξακριβώσουμε επί τη βάση ε, τη διαχείριση και ε, του, του, του, των δομών ελέγχου τι γίνεται με του κινδύνου και με, με αυτού του ελέγχου ε, γίνανε έλεγχοι διαχείρισης και επίσης είχαμε ουσιαστική δοκιμή από τις αρχές ε, του οικονομικού ελέγχου και επίσης ελέγχου επί των δημοσίων διαγωνισμών, διαχείριση επίσης των ε, μέσων ε, δημοσιονομικής διαχείρισης. Κατά τρίτο λόγο που σας είπα, έχουμε ξεκινήσει αυτή τη χρήση των απλουστευμένων εναλλακτικών επιλογών για τις δαπάνες και όσον αφορά τη γεωργία έχουμε τώρα μεγαλύτερο ποσοστό λαθών για την άψη της υπέδρου επίσης και αυτό έχει να κάνει με πάλι την επιλεξιμότητα επίσης ε, τον ΦΠΑ και με μη συμμόρφωση προς εθνικούς κανόνες για να δούμε επίσης το ότι το 2012 το, πρώτο ε, πρόγραμμα σχέδιο δράσης, τα 14 κατημέλη ε, μπήκε σε λειτουργία και οι εθνικές αρχές, οι αρμόδιες ανέφεραν ότι όλα αυτά εφαρμόστηκαν και το 2013. Ε, όλα αυτά τα επεκτείναμε σε όλα τα κρατημέλη. Επίσης έχουμε κάποια κρατημέλη ε, που άλλαξαν τα προγράμματα της υπαίθρου για να ξεκαθαριστούν οι κανόνες που διέπουν τα επιμέρους προγράμματα υποστήριξης. Έχουμε τώρα το κεφάλαιο 7, εξωτερική βοήθεια και έχουμε το καινούργιο στοιχείο τώρα της ε, δειγματοληψίας, το 68% των πληρωμών που έχουν ελεγχθεί, 3,2% όσον αφορά το συνολικό ποσοστό του σφάλματος που είναι 3,3% στο κεφάλαιο 8, έρευνα και άλλες ιστορικές πολιτικές, έχουν 62% των πληρωμών που πέρασαν από έλεγχο και αυτό ε, οδήγησε στο 2,1% του συνολικού ποσοστού σφάλματος, το οποίο είναι 3,9%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερεύνα τώρα τις περιπτώσεις αλλά και τις ε, παρατηρήσεις ε, που έχουν, θέσει, που έχουν τεθεί από το Ελληνικό Συνέδριο για να μην έχουν παρόμοια προβλήματα βράχη πρόθεσμα, μακροπρόθεσμα δε, το ορίζον 2020 πρόκειται να μας οδηγήσει σε περαιτέρω απλούστευση και κατόπιν όλων αυτών των μέτρων για να έχουμε καλύτερες επιδόσεις από τις αρχές των κρατών μελών όπως κατευθυντήριας, κατάρτιση και έλεγχη επιτόπου με συστάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει το καθήκον να προστατεύσει τον προϋπολογισμό με προληπτικά αλλά και διορθωτικά μέτρα η σημείωση 6 που επισυνάπτεται στους ετησίους λογαριασμούς σε σχέση με την πρόσφατη ανακοίνωση για την προστασία του προπολογισμού που προβλέπει να υπάρξει μια γενική υποπτή αυτών των μέτρων αλλά και των επιπτώσεων από πλευράς δημοσιονομικής και να ληφθούν υπόψη ε, η πολυετής διάσταση για τα περισσότερα προγράμματα το 2012 έχουμε και άλλες ε, αποφάσεις ε, διακοπών στα 4,9 δις για ταμεία ε, όπως το περιφερειακό, το Ταμείο Συνοχής, ε, αλληλείας, κοινωνικό και λόγω αυτού του είδους ε, των, των, των δυναμικών ελέγχων φτάσαμε σε αύξηση των ανακτήσεων 4,4 δις το 2012 σε σχέση με το 1,8 το 2011. Ο δε όγκος <clears throat> ή το σύνολο των δημοσιονομικών διορθώσεων και ανεκτήσεων για το περίοδο 9-12 αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε 2% των πληρωμών για την ίδια περίοδο. Όσον αφορά τώρα το Περιφερειακό αλλά και το Κοινωνικό Ταμείο, οι δημοσιονομικές διορθώσει για την περίοδο προγραμματισμού 2006 που τώρα ε, κλείνει, ε, αθρίζεται ή στα 8 δις ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί στο σημαντικό 4% της όλης εισφοράς, η συνεισφοράς των 197 δις. Όσον αφορά τώρα την υγειοργία, οι σορευτικές, οι συνολικές διορθώσεις ε, το, το, των, ε, της εκαθάρισης των λογαριασμών μεταξύ 99 και 12 φτάνουν το 8,3 δις ευρώ και αυτό αντιστοιχεί στο 1,5% των πληρωμών για την ίδια περίοδο. Εάν θεωρείται ότι ο όγκος των διορθώσεων και ανακτήσεων διαχρονικά ε, έχουν έτσι, θα διαπιστώσετε ότι η δυνατότητα διόρθωσης του συστήματος εξασφαλίζει το να έχουμε ένα σημαντικό τμήμα του ποσοστού λάθους που ε, θεωρεί το ελληνικό συνέδριο ότι θα διορθωθεί περισσότερο, θα ανεκτηθεί τα μέσα επόμενα χρόνια και γι' αυτό το λόγο και τώρα να επανέλθω στο πόσο σημαντικές είναι αυτές οι καταποκοπή διορθώσεις που δεν μπορούμε να βρούμε ακριβώς σε ποια ε, σε, ποια από τα κονδύλια που έχουν εκταμιευτεί ε, αντιστοιχούν. Και ακόμα και αν δεν έχουμε άμεσες επιπτώσεις αυτών των διορθώσεων τους τελικούς αποδέκτες και δικαιούχους, ε, αυτά υπάρχει προστασία του προπολογισμού του 2012. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είδε ότι υπάρχουν όσον αφορά κάποια προγράμματα στη Ρωμανία σημαντικά προβλήματα, αλλά δεν μπορούσαμε ακριβώ να δούμε ποιε είναι οι επιπτώσει του και συμφωνήσαμε με τους Ρουμάνους για μια διόρθωση 25% που θα καλύπτει μια δαπάνη ε, η οποία θα αρχίσει να καταλογίζεται από το τέλος του 2012 και από αυτές τις βάσεις η δαπάνη είπαμε ότι ε, αφορούσε παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου και έτσι εξαιρέθηκε από τις ε, δαπάνες και κατόπιν πήγαμε σε κάποιο είδους αντιστάθμιση για την δημοσιονομική διόρθωση οπότε και στην ε, Ρουμανία το Δήμο του 2012 δώσαμε πάρα πολύ λίγα χρήματα αλλά την επόμενη προγραμματική περίοδο ε, είπαμε ότι αν δούμε σημαντικές αντικανονικότητες ως Κομισιόν ή αν βρείτε εσείς αυτό πρόκειται να αφορά τους λογαριασμούς και να τους επηρεάσει όπως τους υποβάλλουν τα κράτη-μέλη και έτσι να έχουμε ε, καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις, οπότε και έτσι θα βελτιώσουμε την κατάσταση στα κρατη στις γεγονές περιπτώσεις όπου έχουμε και αυτές τις αδυναμίες, θα διακόψουν πληρωμές, θα αναστείλουμε προγράμματα και τέλος αυτές οι καθαρές διορθώσεις πρόκειται να βασίζονται σε κάποια αντικειμενικά και κριτήρια διαφάνειας επίση, για να μπορέσουμε να συρρυκνώσουμε τον κίνδυνο για τις δαπάνες της μη επιλέξιμες έχουμε προτείνει να σταματήσει η πρακτική της αναδρομικής χρηματοδότησης και ούτως ώστε κάποιο είδους ελληματικά, προβληματικά προγράμματα θα ε, αντικαθίζονται από κάποια ολοκληρωμένα νέα και επίσης τέλος να σας πω ότι γίνεται όσον αφορά την χρηστή υγιή διαχείριση και επίσης ε, αυτό το, το, το πνεύμα της, ε, ε, το, των, των, επιδόσεων και αποδόσεων διότι εδώ εστιάζεται την προσοχή σας και Είπαμε ότι τώρα θα ξεκινάμε την παροχή περισσότερων πληροφοριών όσον αφορά την προσθέμενη αξία των προγράμματων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τον προϋπολογισμό και περιλαμβάνει και την έκθεση σύνθεσης που βασίζεται στο άρθρο 218 των συνδικών. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντλήσει διδάγματα αυτής της προηγούμενες εμπειρίες και έχει λάβει υπόψη τα, τις προτάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου για την προετοιμασία των προτάσεων της για τη νέα δημοσιονομική περίοδο και όλα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί και από τους νομοθέτες πριν από την έγκρισή τους. Σαφής λοιπόν δείκτες απόδοσης και σαφείς στόχοι είναι τμήματα των προτάσεων της Κομισιόν για το νέο πλαίσιο απόδοσης με τρία σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, ένα σύνολο κυρίων στόχων που πρέπει να επιτευχθούν που συνδέονται με τους στόχους της Ευρώπης 2020. Δεύτερον, περιλαμβάνει δείκτες που αντιμετωπίζουν την προσθέμενη αξία, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και το συνολικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία. Οι διερμηνείς σας ζητάνε να μιλάτε λίγο πιο αργά, λέει ο πρόεδρος. Το τρίτο πλαίσιο απόδοση περιλαμβάνει ε, πρόνοιες για παρακολούθηση και αξιολόγηση ώστε να είναι διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτό θα επιτρέψει μια έγκαιρη απόδοση εκθέσεων σε σχέση με τα αποτελέσματα και την αποδοτικότητα. Το πλαίσιο αυτό θα μας επιτρέψει να καταμετρήσουμε την απόδοση για να αντιμετωπίσουμε τη δύναμα στοιχεία και να βελτιώσουμε την πορεία που θέτουμε. Η Κομισιόν επίσης είναι δεσμευμένη να δημιουργήσει την απαραίτητη αρχιτεκτονική και να υπάρχει καλύτερη καλύτερες έκθεσεις αποδόσεις στο, και καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην έκθεση του άρθρου 318. Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεχίζονται έντονε συζητήσει και προσπάθειε για να υλοποιηθεί αυτό το πλαίσιο. Μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι η Κομισιόν είναι μαζί σα και στη διάθεσή σα για να διευκολύνει τη συζήτηση αυτή που πρέπει να γίνει σε σχέση με την απαλλαγή του οικονομικού έτου 2018. Σα ευχαριστώ τα μάλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιωμέτα, κύριε Επίτροπε, για τις απαντήσεις που δώσατε από την πλευρά τη Κομισιόν. Τώρα έχω ένα μεγάλο αριθμό συναδελφών οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο σε σχέση με την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και σε σχέση με, την, με τα σχόλια της Κομισιόν. Θέλουν να δώσουν σχόλια ή να θέσουν ερωτήσει, αλλά θα δώσω καταρχήν το λόγο στον κύριο Μάρκου Πίπερ. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το μικρόφωνο δουλεύει καλύτερα φαντάζομαι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καλντήρα και τον Επίτροπο κύριο Σιμέτα για τις ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και πληροφοριακές παρεμβάσεις τους και το γεγονός ότι έχουν δείξει διαθεσιμότητα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Εγώ επίσης ε, αναγνωρίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει σημαντικά και αποφασιστικά βήματα. Πρέπει όμως παρόλα αυτά να διαπιστώσω ότι ένα βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι για 19η φορά το ελεκτικό συνέδριο τόνισε πιστοποιητικό αξιοπιστία, συνολικό πιστοποιητικό αξιοπιστία για το 2012 και θα ήθελα επομένω να υπογραμμίσω τέσσερα σημεία σε σχέση με την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου όπου θεωρώ ότι εμφανίζονται τα προβλήματα. Πρώτον, το ποσοστό σφαλμάτων, αυτό καθεαυτό. Δεύτερον, η έκθεση για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει δημοσιευτεί πρόσφατα από την Κομισιόν. Τρίτον, η προετοιμασία για τη συνέχιση της διαδικασίας του, της απαλλαγής του 2011 και τέλος το αποτελεσματόστροφο της ε, στάσης της Κομισιόν που είναι ένα από τα κύρια σημεία που έχουν αναφερθεί. Καταρχήν το θέμα ποσοστό έχει φτάσει από το 3,9% στο 4,8%. Αυτό δεν μας ενθαρρύνει ιδιαίτερα. Είναι για τρίτη χρονιά συνεχής αυτή η αύξηση. Κατανοώ και μπορώ να παραδεχτώ ότι ένα τέτοιο ποσοστό σφαλμάτων και η έλλειψη της ε, δήλωσης αξιοπιστίας πολλές φορές οφείλεται σε πάρα πολλούς κανόνες, σε πάρα πολλές λεπτομέρειες που είναι δύσκολο να τηρηθούν πλήρω. Επομένω είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο να ζητούμε μια τέτοια δήλωση αξιοπιστίας. Και έχουμε και ποικίλου ορισμούς για το τι είδους σφάλματα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά η ίδια η Επιτροπή Μπαρόσο ήταν αυτή η οποία είχε τονίσει ότι θέλει να επιτύχει ένα πιστοποιητικό συνολικής αξιοπιστίας και ότι αυτό θα ήταν ο αντικειμενικός στόχος να επιτευχθεί. Ήταν ο διακεκηρυγμένος στόχος της Επιτροπής Μπαρόσο πριν από μερικά χρόνια, αλλά τώρα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αντίθετα, ανέρχονται συνέχεια τα ποσοστά σφαλμάτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο με λυπεί ιδιαίτερα. Τι, μπορούμε, τι διδάγματα μπορούμε τώρα να <clears throat> αποκομίσουμε. Δεν νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποδηθεί τώρα σε μια συζήτηση σε σχέση με τη μέθοδο το ελεκτικό συνέδριο έχει δικαιολογήσει τη δική του μέθοδο με ισχυρά επιχειρήματα. Η Κομισιόν έχει επίσης παρουσιάσει τη μέθοδο της με ισχυρά επιχειρήματα. Δεν πρόκειται εμείς τώρα να καταλήξουμε σε μια προσπάθεια σύγκρισης ή συγκερασμού των δύο αυτών μεθόδων. Εμείς βλέπουμε ότι έχουμε προβλήματα σε χρονικό επίπεδο πολλές φορές σε ό,τι αφορά την, ε, τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει μια έλλειψη <clears throat> πολλές φορές σημείων εστίασης στη δράση τους και είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς μπορεί να γίνει η συνολική αξιολόγηση αυτών των ενεργειών. Μας ενδιαφέρει όμως να έχουμε καλύτερες πληροφορίες, έχουμε το γεγονός ότι αυξάνονται τα ασφάλματα και η απόλυτη τιμή αυτής της, αυτού του επίπεδου σφαλμάτων ε, και το ποσοστό επίσης οφείλονται στους κλασικούς υπόπτους που είναι τα διαθωτικά ταμεία και τα αγροτικά ταμεία. Επίσης, 60% των σφαλμάτων έχουν ανακαλυφθεί από τα κράτη-μέλη. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Και επίσης, το θέμα της ευθύνη που πρέπει να καταλογιστεί. Εγώ είμαι εδώ και 9 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Γεωργίας έχω δει να συμβαίνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Είναι πάρα πολύ ε, συχνό το πρόβλημα να υπάρχουν προβλήματα στα κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως στις επιδοτήσεις που συνδέονται με τα περιβαλλοντικά θέματα. Αυτό το ξέρουμε και από την έκθεση του κυρίου Γκάιερ. Κάτι όμως το οποίο με εκπλήσει περαιτέρω είναι ότι έχουμε τώρα προβλήματα και στον πρώτο πυλώνα της αγροτικής πολιτικής. Είναι πρόδειλο <clears throat> ότι εκεί υπήρξε η πιο μεγάλη άνοδος και εκεί έχουμε προβλήματα με τον υπολογισμό των αγροτικών εκτάσεων που πολλές φορές παρουσιάζονται λανθασμένα ή ψευδός ε, εκτάσεις αυτού του είδους. Για το ποσοστό σφαλμάτων το πρώτο συμπέρασμα ναι, αυτό το πρώτο, συγγνώμη, το πρώτο συμπέρασμα <clears throat> για τα σφάλματα. Έρχομαι στο δεύτερο θέμα που είναι η έκθεση τη Κομισιόν για την προστασία του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεχομένω θα μπορούσαμε να συνδέσουμε αυτή την ε, θέση τη Κομισιόν με αυτά τα οποία ανέφερε σήμερα το ελεκτικό συνέδριο. Στι 2 Σεπτεμβρίου 2012 η Κομισιόν έδωσε για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια έκθεση για την προστασία του προπολογισμού αυτό ήταν και μια έκκληση του συναδέλφου του κύριου Γκάιερ και θέλω να, τον, το, να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι δεχτήκατε αυτή την έλυση του Κοινοβουλίου και μας δώσατε πολύ σημαντικές πληροφορίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και ληστέλης για μας. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι θα φτάσουν οι πληρωμές στο επίπεδο, φτάσαν τα, στο 14 ε, δισεκατομμύρια ευρώ, 4,4 ήταν το ποσοστό σφαλμάτων και αν συνυπολογίσουμε όλους τους, ε, ε, όλες τις διορθώσεις έχουμε διορθώσει για 3,2% των συνολικών πληρωμών. Εδώ όμως πρέπει να θέσω ένα ερώτημα. Είπαμε ότι πρόκειται για 4,4 δισεκατομμύρια τα οποία υφίστανται, υπέστησαν μάλλον διορθώσεις Πόσα από αυτά τα 4,4 δισεκατομμύρια ανακτήθηκαν και επανήλθαν στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Ή πόσο θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία διόρθωσης. Ποιο είναι το διοικητικό κόστος και άχθος για να μπορέσει να γίνει αυτή η διόρθωση. Τι απώλειες τόκων υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν χρήματα τα οποία παρέμειναν εν αδρανία δεν χρησιμοποιήθηκαν. Και αυτό είναι και επιπλέον ε, φόρτος για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Προφανώς αυτό δεν είναι σφάλμα της Κομισιόν, είναι απλώς οι πρόνοιες που βρισκόνται σε ορισμένου κανονισμούς, είτε μέχρι το 2006 είτε από το 2007 και επέκεινα, που επέτρεψαν στα κράτη-μέλη να αντικαταστήσουν προβλήμα, προγράμματα τα οποία ήταν προβληματικά, να τα αντικαταστήσουν με νέα προγράμματα. Δεν υπάρχει όμως καμία εγγύηση ότι τα νέα αυτά σχέδια και προγράμματα στα κράτη-μέλη οδήγησαν σε βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας. Αντίθετα, φαίνεται ότι τα νέα προγράμματα αυτά παρουσίασαν τα ίδια σφάλματα όπως και τα παλαιότερα προγράμματα. Είναι αξιοσημείωτο 58% των ε, ε, κοινής διαχείρισης προγραμμάτων σε ένα κράτος μέλος ε, δεν εκτελέστηκαν. Πρόκειται για την Ισπανία. Και στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα μόνο τρία κράτη-μέλη ήταν αυτά. Τα, υπήρξαν τρία κράτη-μέλη που ήταν υπεύθυνα για 80% των σφαλμάτων Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ανήκει μόνο στο παρελθόν. Και οι στατιστικέ τη κομισιόν δείχνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Είναι οι χώρε με το υψηλότερο ποσοστό σφαλμάτων και ακολουθεί η Τσεχία, η Πολωνία και η Ρουμανία. Μπορούμε να δούμε λοιπόν με σαφήνεια ότι υπάρχουν προβλήματα με τα αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι ένα φαινόμενο που συνεχίζεται εδώ και χρόνια ή δεκαετίες. 60% των σφαλμάτων που υπόκειται στην κοινή διαχείριση θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί αν τα κρατημέλη είχαν κάνει σωστά το έργο τους. Τι συμπέρασμα λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε από όλα αυτά. Και επίσης μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής μας ήρθαμε σε επαφή με τον Ισπανό Υπουργό, ο οποίος είναι αρμόδιο και ζητήσαμε να έλθει ενώπιον τη Επιτροπή μας και επίση ο κύριο Γκάιερ είχε οργανώσει μία συνάντηση με τον Τσέχο και Ρουμάνο αρμόδιο Υπουργό και θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη του Ισπανού Υπουργού για τα ίδια θέματα αυτά. Είναι φανερό λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη έχουν κάνει σημαντικές παραλήψεις. Αλλά το γεγονό ότι διαρκεί αυτή η διαδικασία εδώ και δεκαετίε, δύο δεκαετίε, θα πρέπει η Κομισιόν να λάβει υπόψη τη πιο σοβαρά το ρόλο τη ω θεματοφύλακα των συνθηκών. Το να μπορούμε να αλλάσουμε συνέχεια προγράμματα και σχέδια μέχρι να μπορούν να τύχουν επιδοτήσεων και με τον τρόπο αυτό να παραβιάσουμε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής αυτό πρέπει να σταματήσει. Να το πω πάρα πολύ Σαφώς. Άμα έχουμε κάποιον ο οποίος κάνει συνέχεια οδικές παραβάσεις με τον ίδιο τρόπο, κάποια στιγμή θα πρέπει να του πάρουμε και το δίπλωμα. Ενώ αυτό βέβαια δεν βλέπουμε να γίνεται με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε λοιπόν με τα περιφερειακά προγράμματα. Εάν δεν λοιπόν ικανοποιεί κανείς τους κανόνες, δεν μπορεί να παίρνει συνέχεια καινούρια προγράμματα. Δεν μπορεί κανείς να λέει ότι όταν κάνεις ε, παραβάσεις θα σου δώσω ένα καινούριο αυτοκίνητο για να μην κάνει παραβάσεις. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αλλάζει τα πράγματα. Δεν μπορούμε με τον τρόπο αυτό να αλλάξουμε την κατάσταση στα επίπεδα του προπολογισμού, αν δίνουμε πάντα νέο χρήμα σε αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει κακοδιαχείριση των προηγουμένων κονδυλίων. Γι' αυτό εγώ ζητώ να υπάρξει άντληση συμπερασμάτων για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Χρειαζόμαστε, όπως είπε και ο Επίτροπος κ. Σεμέτα, χρειαζόμαστε να υπάρξει κάποιος αυτόματος μηχανισμός ο οποίος θα επιφέρει χρηματοδοτικές διορθώσεις. Δηλαδή τα κάτι μέλη που έχουν υψηλό ποσοστό ε, σφαλμάτων θα πρέπει να υφίστανται μια ιδιαίτερη εποπτεία. Μπορεί να υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία όπου σε, σε, συνάρτηση με τα, το ποσοστό σφαλμάτων θα υπάρχει ισχυρότερη εποπτεία και έρευνα από την Κομισιόν. Οι χώρες που έχουν μεγαλύτερο ποσοστό θα έχουν μεγαλύτερο έλεγχο από την Κομισιόν. <clears throat> Νομίζω με το να υπάρξει μια τέτοια πιο αυτόματη διαδικασία θα μπορέσουν να αλλάξουν τα πράγματα. Βέβαια, θα πρέπει να πιστούν και οι συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αρμόδια επιτροπή για τα θέματα αυτά. Δεύτερον, τώρα έχω να κάνω μια πρόταση στο ελεκτικό συνέδριο, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από το ελεκτικό συνέδριο στις εκθέσεις του κατά χώρα να αναφέρει και τα αίτια, γιατί πάντα είναι οι ίδιες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό σφαλμάτων. Και σε ό,τι αφορά το θέμα των συνθήκων. Γιατί δεν πρέπει το ελεκτικό συνέδριο να εξειδικεύει ανακράτος μέλος αυτά τα οποία περιέχει η έκθεσή του. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, δεν υπάρχει κάποιο άρθρο των συνδικών που το απαγορεύει. Αυτό νομίζω το ελεκτικό συνέδριο έχει κάθε υποχρέωση να ελέγξει καλύτερα τα σφάλματα αυτά. Όταν βλέπουμε ότι είναι ορισμένε περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπου συγκεντρώνονται τα 80% των σφάλματων, είναι υποχρέωση και του ελεκτικού συνεδρίου να ελέγξει καλύτερα τα πράγματα αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει και ζητώ λοιπόν και από το ελεκτικό συνέδριο να σκεφτεί καλύτερα για το θέμα αυτό. Εξέφρασα στην αρχή μου τις ευχαριστίες, στην αρχή της ευχαριστίας μου για το ελεκτικό συνέδριο για όλα αυτά τα νέα στοιχεία που μας έχει δώσει σε ένα σημείο όμως πρέπει να εκφράσω την εμβροντισία μου, διότι στην πρόσφατη έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, στην σύντομη ε, επίτομη ε, έκδοση που αφορά τους πολιτικούς και τους ε, δημοσιογράφους, αναφερθήκατε σελίδα 7 στη δήλωση αξιοπιστίας, όπου σε μισή σελίδα αιτιολογείται γιατί δίνεται μια αρνητική ε, δήλωση αξιοπιστίας ή μάλλον δεν μπορείτε να δώσετε μια θετική δήλωση αξιοπιστίας. Μα σε ένα χρόνο που ανεβαίνουν ε, όπου αυξάνονται τα σφάλματα, γιατί δεν υπάρχει μια τέτοια αρνητική αιτιολόγηση στο σύντομο κείμενο που είναι για τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς, αλλά μόνο στο μεγάλο κείμενο βλέπω αυτή η αναφορά για τα αρνητικά αποτελέσματα αυτά να βρίσκεται μονάχα, ψάχνω τώρα να βρω την, τη σελίδα. Μα δεν τη βρίσκω κιόλα. Κάπου λέτε γιατί καταλήξατε σε, αρνητική γνώμη για την αξιοπιστία, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι επαρκής αιτιολόγηση. Σελίδα 5 λοιπόν. Στο σκιασμένο, γραμμοσκιασμένο κείμενο περιγράφεται κάτι το οποίο στην προηγούμενη έκδοση κάλυπτε μια ολόκληρη σελίδα. Αυτό είναι ένα κέριο σημείο της έκθεσής σας. Σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να μην είναι συγκεκαλυμμένα αυτά τα στοιχεία που έχετε, εάν έχετε να πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, να το πείτε. Δεν θεωρώ ότι είναι σημεία τα οποία πρέπει να αποκρύπτονται. Τρίτο σημείο, και πάω και πιο γρήγορα λιγάκι, η ευθύνη της Κομισιόν σε σχέση με τη συνέχεια που δίνεται στην έκθεση Γκάιερ, δηλαδή για την έκθεση απαλλαγής του 2011. Η Κομισιόν έχει δράσει για δύο εκκλήσεις του Κοινοβουλίου. Καταρχήν η ανακοίνωση για την προστασία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και δεύτερον για το άρθρο 318 που αφορά τις αξιολογήσεις. <clears throat> Μια μεγαλύτερη στατιστική διαφάνεια είναι κάτι το οποίο εμείς το αναγνωρίζουμε και το χαιρετίζουμε. Αλλά δεν έχουμε ακόμα κατά την άποψή μας τα απαραίτητα μέτρα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση και εδώ νομίζω ότι αντανακλώ και αυτό το οποίο λέει ο κύριος Γκάιερ, ότι δεν βρήκαμε κάποιες καινούργιες προτάσεις. Οι ελλείψεις που βρέθηκαν στο πρώτο πυλώνα της αγροτικής πολιτικής εξακολουθούν να είναι ακριβώς οι ίδιες όπως και πέρσι. Απλώς και μόνο αυξάνει το ποσοστό δυστυχώς των σφαλμάτων σε ό,τι αφορά την αγροτική ανάπτυξη. Βλέπουμε και πάλι τα ίδια επιχειρήματα να αναφέρει η Κομισιόν όπως και πέρσι και λαμβάνει υπόψη και μια ε, ένα σχόλιο του Συμβουλίου του, του, του, της 29ης Νοεμβρίου 2012 αυξάνει και εκεί το ποσοστό σφαλμάτων για το χρηματοδοτικό εργαλείο στην πολιτική συνοχής η Κομισιόν δεν μας δίνει τίποτα νέο από αυτά που είχε αναφέρει το Φεβρουάριο του 2012 για την τότε απαλλαγή. Η Κομισιόν λοιπόν επαναλαμβάνει τα ίδια αλλά δεν έχει αντιμετωπίσει το γεγονός ότι τα ασφάλματα αυτά εστιάζονται σε λίγες μονάχα χώρες μέλη. Ζητώ λοιπόν από την Κομισιόν να υπάρξουν νέα, νέες ενέργειες για τα θέματα αυτά. Να σταματήσει λοιπόν η Κομισιόν να πετάει σε άλλους το μπαλάκι. Δεν γίνεται να συνεχίσει αυτή η διαδικασία. Θέλω να ζητήσω λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει απαλλαγή μονάχα στην περίπτωση που η Κομισιόν δέχεται στο μέλλον να δημιουργήσει μηχανισμούς αυτόματης διόρθωσης που θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο. Μια τελευταία παρατήρηση σε ό,τι αφορά την καταμέτρηση της ε, απόδοσης. Αυτό φαίνεται για πολλούς ότι είναι σημαντικό, πρέπει να προσθεθεί στη διαδικασία της απαλλαγής και αναφέρεται και σε αυτό και η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Πρέπει όμως να σας πω ειλικρινά ότι δεν θεωρώ ότι είναι επαρκώς σαφής η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία αυτού του εγχειρήματο. Και αυτά που κάνει η Κομισιόν και το Ελεκτικό Συνέδριο όσο προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταμετρήσει καλύτερα τις ε, επιπτώσεις στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, τόσο περισσότερο βρισκόμαστε σε σύγκρουση με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Θα πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα πού τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν κάτι το οποίο αποτελεί επίτευξη ευρωπαϊκών στόχων και δεν αντικαθιστούν τα εθνικά κονδύλια. Δεν μπορούμε <clears throat> να συνεχίσουμε να παίζουμε. Το θέμα είναι, σαν να είμαστε μικρά παιδιά, το θέμα είναι να δούμε πού υπάρχει πραγματικά μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και αυτό είναι σημαντικό εν ώψη και της στρατηγικής Ευρώπης 2020. Μα ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε περισσότερε υποδομέ, να βελτιώσουμε την επαγγελματική κατάρτιση στην Ευρώπη. Αυτά είναι παραδείγματα ε, για την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Όλα αυτά τα οποία λέγονται για προσωπικούς δείκτες σε ό,τι αφορά την προσωπική ανάπτυξη και όλα αυτά, αυτό είναι ένα διέξοδο για μένα. Δεν είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταμετρήσουμε την πρόοδο στο κοινωνικό επίπεδο. Μόνο με τη δημιουργία δομών μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και όχι με καταποκοπήν ή σε ατομικό επίπεδο δείκτες. Κυρίε και κύριοι, λοιπόν, <clears throat> ποια είναι τα συμπεράσματά μου. Η διαδικασία απαλλαγή έχει μόλις ξεκινήσει. Θα ήθελα να συνεχίσει μία διαδικασία ερωτήσεων προς το Ελεκτικό Συνέδριο και την Κομισιόν και διατύπωσης αιτήσεων από, το, από την πλευρά του Κοινοβουλίου και μία πρώτη αίτηση είναι ότι η Κομισιόν πρέπει να δείξει μεγαλύτερη ενεργητικότητα σε ορισμένου τομεί, του οποίου κατονόμασα και απαρίθμησα προηγουμένω. Εγώ σα είπα προηγουμένω τι μπορεί να κάνει κανεί για τα θέματα αυτά. Και δεν θέλουμε απλώς ε, υπεκφυγές ή ελιγμούς αποφυγής περιμένω και από την Κομισιόν και από το Ελεκτικό Συνέδριο να δείξουν πνεύμα συνεργασίας και θέλω επίσης να παροτρύνω και τους συναδέλφους μας να συμμετάσχουν στη συζήτηση με το Ελεκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή για το θέμα αυτό και να θέσουν ε, ερωτήματα κριτικού χαρακτήρα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα που μας απασχολεί. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος, τον Μάρκους Πίπα και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στις πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι είναι 10 αυτοί οι οποίοι έχουν ζητήσει να λάβουν το λόγο. Ο πρόεδρος του ελεκτικού συνεδρίου σας <clears throat> υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να φύγει στις 11. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Θα ήθελα να δώσω λοιπόν στους συντονιστές ή τουλάχιστον σε ένα εκπρόσωπο κάθε πολιτικής ομάδος και μετά θα μπορούσαν να λάβουν το λόγο ή τα υπόλοιπα μέλη των κομμάτων με σύντομες παρεμβάσεις ενός ή ενάμιση λεπτών. Παρακαλώ, ο Ντέρεκ Ουάν. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και το ελεκτικό συνέδριο για την έκθεσή του και την αρχική απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως και ο μας το όλοι απογοητευμένοι διότι αυξήθηκε προς το σφαλμάτων από 3,9% στο 4,8%. Κάθε χρόνο από το 2009 και μετά είχαμε αύξηση στο ποσοστό σφαλμάτων. Και κάτι άλλο που με απογοήτευσε και τα συζητήσαμε αυτά. Είναι ότι αυτό δίνει πυρομαχικά και σκεπτικιστές στα κράτη-μέλη. Να πω στους συναδέλφους ότι βλέπουμε τίτλους σε κάποιες βρετανικές εφημερίδες σύμφωνα οποίες ε, δεν λειτουργεί σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λαμβάνουν, ότι κάνει απάτες, δεν λαμβάνουν υπόψη τη διαφορά μεταξύ σφαλμάτων ε, και απατών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δύσκολη η χαλεπή οικονομική καιρή, άρα πρέπει να δαπανάτε σωστά κάθε ευρώ και έγκαιρα. Να δημιουργεί θέσει απασχόλησης και ανάπτυξης σε κάθε κάτω και σε κάθε περιφέρεια. Γι' αυτό εγώ θέλω στην έκθεση να δω ποιοι είναι οι λόγοι για την ύπαρξη των σφαλμάτων. Γιατί αυξήθηκε το ποσοστό των σφαλμάτων. Θέλω να δω τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον για να μειωθεί το ποσοστό σφάλματο στι δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε την έκθεση του λεκτικού Συνεδρίου, βλέπει κανεί ότι σε κάθε κεφάλαιο, σε κάθε τμήμα αυξάνεται το ποσοστό σφαλμάτων και κάθε επίτροπος θα έχει εξήγηση για την αύξηση αυτή και για κάθε τμήμα. Η Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση θα πει ότι 14% της αύξησης οφείλεται σε μια χώρα, στη Ρουμανία. Και χωρίς αυτό η πραγματική αύξηση στη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση θα ήταν λιγότερο από 2%. Κάθε επίτροπος θα έχει δικαιολογία για την αύξηση. Σήμερα εγώ θα ήθελα να δούμε κάποια από τα γενικότερα ζητήματα τους γενικότερους λόγους που δίδονται για τη γενική αύξηση των σφαλμάτων. Πρώτον, αλλάζουν οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί το ελεκτικό συνέδριο. Η δειγματοληψία έχει αλλάξει. Το ελεκτικό συνέδριο στην έκθεσή του φρονεί ότι 0,3% της αυξήσεως οφείλεται στη μεθοδολογική αλλαγή. Και ο πρόεδρος του ελεκτικού συνεδρίου εξήγησε τις υιοθετηθήσεις αλλαγές για το 2012. Τακτικές αλλαγές όμως στη μέθοδο δεν είναι κάτι επικοδομητικό, αυτό πιστεύω εγώ. Το λέκτικό συνέδριο μπορεί να μας πει αν προτίθεται να κάνει μεθοδολογικές αλλαγές στο μέλλον, κάτι που μπορεί και πάλι να επηρεάσει το ποσοστό σφαλμάτων. Δεύτερον, κάτι που είπαν αρκετοί επίτροποι και αξιωματούχοι. Το λεκτικό συνέδριο μετά τα σφάλματα ακόμα και όταν κατά αποκοπήν οικονομικές διορθώσεις έχουν λάβει χώρα. Ο Επίτροπος το είπε αυτό στην παρέμβασή του. Ερώτηση για το εθνικό συνέδριο. Δέχεστε ότι όταν έχουν γίνει διορθώσεις ότι ο προπολογισμό Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχει προστατευτεί και αν αυτό είναι δεκτό αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην έκθεση. Τρίτον, πάντα το συζητούμε αυτό στην Επιτροπή. Όταν συζητούμε κυρίω την ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Δηλαδή, ποιο είναι ο λόγο των κρατών μελών. Δεν αποτελεί μυστικό ότι λίγα κάτι μέλη δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα και ο εισηγητή στην παρέμβασή του κατανόμασε κάποια κάτι μέλη. Υπάρχουν και ζητήματα και προβλήματα σε άλλα κάτι μέλη όμω. Στον Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματι, οι πληρωμέ των διεθντικών ταμείων έχουν ανασταλεί. Δεν είναι προβληματικά τα κάτι μέλη που ανέφερε ο εισηγητή, αλλά εμπλέκονται και άλλα κάτι μέλη. Και τα προβλήματα των κατών μελών συμπεριλαμβάνουμε του κανόνε δημοσίων προμηθειών ε, διάφορες προσεγγίσεις ανθασμένες, τα ελεγκτικά συστήματα που δεν εντοπίζουν ή δεν εμποδίζουν την διάπραξη σφαλμάτων. Πέρσι ο Γιάνν Σκέιερ στην έκθεσή του εκτίμησε ότι 62% των σφαλμάτων θα μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί από τα κράτη-μέλη. Η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου αυτό το επιβεβαιώνει εκ νέου. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προσπαθήσει να βρει ένα μηχανισμό ο οποίος θα εντοπίζει καλύτερα τα προβληματικά κράτη-μέλη σε έγκαιρο στάδιο, να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για να μειώνονται τα σφάλματα και χρειάζεται καλύτερο σύστημα για διακοπές και αναστολές και διορθώσεις στις πληρωμές. Ο εισηγητής επιθυμεί διακαώς αυτό να το εξετάσει, το συζητήσαμε αυτό. Δηλαδή να θεσπίσουμε κάποιο μηχανισμό που θα δημιουργεί ένα πολύ ε, στέρεο σύστημα στο μέλλον. Και κάτι άλλο. Ο πρόεδρος του λεκτικού Συνεδρίου έκανε ένα σχόλιο. Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προετοιμάσει μια θέση μακροπρόθεση όσον αφορά την ε, ροή, την οικονομική των, ε, του ρευστού. Δύσκολο αυτό να προγραμματιστεί. Θέλω κάποιες πληροφορίε από αυτού. Έκανε πρόβλεψη ο πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου για επιδόσεις. Ευπρόσδεκτο αυτό. Στο νέο γύρο προγραμμάτων οι επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε σχέση με τις δαπάνες πρέπει να βελτιωθούν. Αν δείτε τους σχετικούς κανονισμούς για τα επόμενα προγράμματα, γίνονται σχετικές προτάσεις για να προβλέπονται μελλοντικές επιδόσεις. Θα συζητήσουμε τις επιδόσεις, την ερεσιμότητα, αποθεματικά, θεματική συγκέντρωση στα περιφερειακά ταμεία. Λοιπόν, θα έχουμε καλύτερες προβλέψεις να αφορά τις επιδόσεις στο μέλλον. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα εστιαστούμε καλύτερα σε επιδόσεις στο μέλλον. Θα μπορέσουμε να προσμετρήσουμε τις επιδόσεις στα επόμενα προγράμματα. Γιατί αυτό θα είναι κλειδί. Τέλος. Συμφωνώ με τον πρώτο του ελεκτικού συνεδρίου. Είπε, κλείνοντας, ότι θεωρούσε ότι είναι σημαντικό να συνεργαστούμε για τα θέματα αυτά. Κατά την άποψη της ομάδας μας θέλουμε να συνεργαστούμε με τους πάντες. Έτσι στο μέλλον τα ποσοστά σφαλμάτων του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκής Ενωση θα μειωθούν και θα χρησιμοποιούμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεσματικότερα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος και επόμενη είναι η κυρία Γκρέσλη και κατόπιν ο κύριος Μίλλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά αυτά τα οποία μας παρουσιάσατε της έκθεσης και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο 1 ήδη ετέθηκαν κάποια ερωτήματα και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποια ερωτήματα για το ποσοστό σφαλμάτων. Έχω την εντύπωση μετά από αυτά που αναφέρατε ότι ο έλεγχος των ελέγχων έχει σταθεί αποτελεσματικός. Αλλά λέτε ότι στα διαστατικά ταμεία 50% των σφαλμάτων δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και επομένως δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει το σύνολο των ζημιών που προέρχονται. 50% είναι πολύ. Εγώ νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά με τη μέθοδο που ακολουθήθηκε. Και όλα αυτά τα οποία αναφέρονται την εντύπωση ότι υπάρχει ενδεχομένως και κάποια χειραγώγηση του ποσοστού των σφαλμάτων. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και τα έχει αναφέρει και ο συγητής της Επιτροπής μας. Εγώ δεν ε, <clears throat> θεωρώ ότι υπάρχει σωστή προστασία των ε, οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν περνάνε στους εθνικούς προϋπολογισμούς ε, κονδύλια τα οποία δεν θα έπρεπε να δίδονται βάσει των δημοσιονομικών κανονισμών. Το ευρώ του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διαφέρει από ένα ευρώ εθνικού προϋπολογισμού. Όταν έχουμε ένα τόσο προβληματικό πλαίσιο δεν έχει νόημα να λέει ένα κράτος μέλος ότι εγώ θα καλύψω το δικό μου <clears throat> τμήμα των ε, σφαλμάτων και δεν με ενδιαφέρει το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι τα, οι φορείς πιστοποίησης δίδουν συστηματικά λανθασμένες πιστοποίησεις, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει η Κομισιόν να το αντιμετωπίσει όλα αυτά τα μέτρα που έχουν λάβει τα κρατημέλη δεν έχουν οδηγήσει σε καλύτερο επίπεδο και υπάρχουν ακόμα και συγκρούσεις συμφερόντων μέσα στα κρατημέλη. Προφανώς δεν θέλουν να πούν ότι υπήρξε λανθασμένη χρήση κονδυλίων, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε πρόστιμα για αυτούς. Αν τα κρατημέλη λοιπόν <clears throat> ε, ανακαλύπτουν τα ασφάλματα, θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία που να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να κρατάνε τα χρήματα αυτά. Παρ' όλα αυτά, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο μεγάλα προβλήματα με τους φορείς πιστοποίησης και εδώ κύριε Πρόεδρε του Ελεκτικού Συνεδρίου θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη διευκρίνηση. Νιώθω κάποια λοιπόν απογοήτευση γιατί είναι η τρίτη χρονιά που ανεβαίνουν τα ποσοστά ασφαλμάτων. Θα ήθελα λοιπόν εδώ πέρα να υπάρξει μια σαφέστερη εξήγηση γιατί συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και έχουμε επίσης και αλλαγές στα κράτη-μέλη, ε, λόγω της κρίσης έχουν διακοπεί κάποια προγράμματα και σε κάποια κράτη-μέλη λόγω της κρίσης έχουμε φτάσει σε 95% χρηματοδότηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν συμμετέχουν τα κράτη-μέλη. Στις περιπτώσεις λοιπόν που υπάρχει ένα σφάλμα, μήπως θα πρέπει να φροντίσουμε να διορθωθούν τα πράγματα ε, αμέσως, γιατί δεν έχουμε και πολλά χρήματα να δώσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο κύριος μιλτερ και ο κύριος Στάς Ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο του Λεπτικού Συνεδρίου που μας παρουσίασε την έκθεση. Μία από τα ίδια είναι πάνω κάτω. Εγώ ήλπισα ότι ως βουλευτής κάποια στιγμή θα είχα την εμπειρία ενό θετικού ντάς. Αλλά από ό,τι φάνηκε ήταν αυτά φρούδες ελπίδες. Μεγάλη απογοήτευση. Αλλά ακόμα πιο μεγάλη είναι ότι όλα τα στοιχεία, τα αριθμητικά είναι από πριν. Ακόμα και για τη Γεωργία το ποσοστό του λάθους ήμασταν στο 2% και τώρα είμαστε στο 3,8% τουλάχιστον αυτά λέει η έκθεση για πρώτη φορά σήμερα το πρωί το είδα άρα τι γίνεται ποιος είναι ο κίνδυνος που ελοχεύει διπλασιασμό του σφάλματος περίπου σε ένα λάθος ανάπτυξη της υπαίθρου, περιφερειακή πολιτική κλπ Παντού, παντού το σφάλμα είναι πολύ ψηλά. Και τα κράτη-μέλη βεβαίως είναι ο βασικός ένοχος. Για άλλη μια φορά σας τονίζω ότι πρέπει να πιέσουμε. Ευτυχώ είναι στο πλάνο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάμε κάτι να αποσπάσουμε κάτι μέλη σαν δήλωση, τώρα και κάτι άλλο. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν ο σημερινός πρόεδρος της Κομισιόν ανέλαβε τα καθήκοντά του και θυμάμαι ότι και τότε ήταν ταραγμένη η και είχε πει ότι σε πέντε χρόνια θα έχουμε θετικό ντάς. Διακόπηκε ο Σμίλτερ. Τι να σας πω. Δεν ξέρω ποια πενταετία ενώσε. Τώρα είμαστε εννιά χρόνια μετά. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μα εξηγήσει ο πρόεδρο γιατί πριν από 9 χρόνια ήταν τόσο αισιόδοξο. Τι να πούμε. Κάθε χρόνο επί οικής προς την Κομισιόν αναβάλουμε, θεωρούμε, ελπίζουμε ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα παρά το ότι όλα σα γίνονται είναι κόντρα στις υποσχέσεις. τας, τι πιθανότητες έχουμε, δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει καν το, σύστημα αυτό του υπολογισμού. Τι γίνεται. Για τον προηγούμενο υπολογισμό πόσο του σφάλματος δεν υπήρχε καμία διαμαρτυρία, κανένα παράπονο. Γιατί άλλαξε τότε, ας μου πει κάποιο. Κατά τα λοιπά, σε αυτή τη φάση ας μελετήσουμε την έκθεση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πάντως, εν των εκλογών θα είναι δύσκολο. Να προσπαθήσουμε να δείξουμε σοβαρότητα, να αφήσουμε κάποια προοπτική ότι κάτι θα γίνει. Δεν φταίει το ελεύθερο συνέδριο. Ανέκαθεν το σεβόμουν όμως έχει αρχίσει να κλονίζεται αυτή μου η εκτίμηση και ο σεβασμός. Και δεν φταίει καθ' αυτό το ελληνικό συνέδριο. Φταίει το Συμβούλιο. Μην κρίναμε τον Τάσο. Αλλά είδατε τι έγινε με το μέλος από την Κροατία. Αυτό ήταν ανοιχτός πόλεμος και τελικά στιγματίστηκε και μαυρώθηκε το ελληνικό συνέδριο. Εμείς πάντως ακόμα δεν έχουμε θεωρήσει ότι έληξε η υπόθεση εκείνη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τέτοια πράγματα. Δυστυχώς η Ιωνή είναι δυσάρεστη και θα πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Μπάρτης, ο επόμενος ομιλητής. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όσον αφορά αυτά που ακούσαμε τώρα από τον Γιάν Μίλτερ, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Τα, συ, συζητήσαμε χθε το απόγευμα με το υποψήφιο μέλος. Κύριε Καλτέρα, αυτό πρόκειται να είναι ένας λεκές που θα αμαυρώνει την υπηρεσία σας και δεν φταίνει οι συνάδελφοί σας και εσείς. Αλλά φταίει το πρόσωπο εκείνο το οποίο δεν έλαβε υπόψη τι ευαισθήσει το κοινοβούλιο και πώς λειτουργεί ένα κοινοβούλιο. Αλλά φταίει το Συμβούλιο που προχώρησε ή στον ορισμό, καθορισμό αυτής της ε, υποψηφιότητα. Τέλο πάντων, ευχαριστούμε όσον αφορά την ετησία και ευχαριστούμε όλου του επιμέρου του ε, συναδέλφου σα και τον προσωπικό σα γιατί το έργο που επιτελείται είναι πάρα πολύ αξιόλογο. Μας ε, δίνεται τόσες και τόσες πληροφορίες. Και εμείς, για να δούμε, τι θα κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες. Ξέρω ότι δεν θα κάνουμε, θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητούμε περί της μεθόδου. Δεν έχει νόημα αυτό. Δεν είναι αυτό το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε προς τα έξω. Με τι έχει νόημα, τι έχει σημασία. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία πρέπει να σας τονίσω ναι, και υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες συγκεκριμένες με και με αυτό το οποίο κάνετε θα πρέπει ξεκάθαρα να το πούμε. Τι γίνεται όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική, την ενέργεια, τη γεωργία. Πάνε στο 42% των κονδυλίων και <coughs> είχαμε πει το 25% των δαπανών της γεωργίας θα μπορούσε να λυθεί από τα κράτη-μέλη για την ελευθερική πολιτική 18%, για την περιφερειακή πολιτική 56%. Τις πληροφορίες τις είχαν τα κρατημέλη, μπορούσαν κάτι να κάνουν. 6% για, για κοινωνική πολιτική. Ξέραμε, ξέραμε το, το, το του λάθους. Αυτά ήταν πόστο του λάθους. Το ξέραν τα κρατημέλη. Και δεν μιλούμε τώρα για απάτη. Μιλούμε για ανακριβείς καταχωρήσεις οπότε και τα κρατημέλη είχαν τα στοιχεία που έπρεπε και έτσι μπορούσαν να κάνουν κάτι. Πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Κύριος Πίπερ, έκανε μια σύγκριση μεταξύ αυτών των σφαλμάτων και των τροχαίων παραβάσεων και πώς κανείς Άμα το παρακάνει μπορεί να φτάσει να του πάρει το λομαδίγηση. Κύριε Καλτέρα, στη σελίδα 11 κάτι λέτε εκεί για τις δημοσιονομικές διορθώσεις και εκεί αναφέρεται τα κράτη-μέλη στις περισσότερες των περιπτώσεων συμφωνούν με τις διορθώσεις αυτές. Όμως, στη συνέχεια, τι λέτε. Λέει στα αγγλικά αυτό, αυτά πρόκειται να γραφούν ε, σε άλλα κονδύλια Οπότε και τελικά εδώ σημειώνεται συμφωνία όσον αφορά τις δημοσιονομικές διορθώσεις. Μιλούμε για αυτά τα χρήματα τα οποία πλέον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω των διορθώσεων, αλλά θα συνεχίσει να τα έχει το σχετικό κράτος μέλος να τα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει μια κλίση διατροχή παράβαση και ταυτόχρονα παίρνει τα ίδια χρήματα και πάει στους μάρκετ να ψωνίσει. Κάποια κράτη-μέλη ευθύνεται για το είπαμε για το 80% των σφαλμάτων, το είπε ο συγκεκριτή ξεκάθαρα και οπότε κύριε Επίτροπε θα πρέπει να κάνετε και να καταστρώσετε κάποιο σχέδιο. Μιλούμε για την περίοδο 14-20. Καθίστε και σκεφτείτε ένα σχέδιο. Πώς για εκείνα τα κράτη-μέλη που είπαμε ότι ξέρουν σε 90 τόσο τις τι συμβαίνει. Βέβαια υπάρχουν κάποια λίγα κράτη που δεν έχουν ελεγκτικούς μηχανισμούς, δεν ασκούν ελέγχους. Άρα εσείς καθίστε να δείτε τι θα τα κάνουν αυτά τα κρατημέρια για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε. Θα σταματήσουν αυτή την πρακτική και κάτι θα κάνουν. Να ανασταλούν πληρωμές και εκταμιεύσεις αν χρειάζεται. Και είδαμε τι έγινε με τη γεωργία στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Αναστήλαμε πληρωμές και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα βελτιώσεις. Αυτά όλα καταστούν προϋποθέσεις απαλλαγής. Επίσης, σε αυτή τη διαδικασία της απαλλαγής θα πρέπει να δούμε πώς θα κάτσουμε και θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα δράσης. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αποτελεί τον κόδρα του κινδύνου που κρούεται. Θα πρέπει πάντως να κάτσουμε να βρούμε και κάποιο είδου γενικότερο σχέδιο να συνεργαστούμε. Όλα τα θεσμικά όργανα προς τούτο. Πρόεδρε, κατά αυτή τη διαδικασία της απαλλαγής, τι διαπιστώνουμε, ότι δεν μας παίρνει στα σοβαρά το Συμβούλιο. Τι κάνουμε, κάτι καλύπτει ο ένας τον άλλο. Άρα, ας πούμε στο Συμβούλιο να μας πάρει σοβαρά, να σταματήσουμε να καλύπτουμε ο ένας τον άλλο και σε συνεργασία με τον εισηγητή, τους σκιώδες, ό, η Επιτροπή μας, όλο το Κοινοβούλιο να κάτσει να φτιάξει ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο και να καλύψουμε όλα αυτά που μας έχει επισημάνει το Ελληνικό Συνέδριο τα τελευταία 19 χρόνια. Όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη και να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα δράσης. Και έτσι να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το 91% των σφαλμάτων τα οποία μπορούσαν να τα έχουν λάβει υπόψη τα κράτη-μέλη θα αποτελεί παρελθόν. Να τα κάνουμε όλα αυτά τους αμέσως επόμενους μήνες. Αυτό θα πρέπει να γίνει, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Άσεν για την ε, ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. I would like to... Θα ήθελα ρωτήσω το ελεκτικό συνέδριο. Συμφωνούν με τις δικαιολογίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση των σφαλμάτων στο 4,8%. Λένε ότι αυτό οφείλεται στην αλλαγή τη δειγματοληψία από πλευρά ελεκτικού συνεδρίου. Διαβάζοντα την έκθεση, βλέπω ότι το ελεκτικό συνέδριο το ίδιο αναγνωρίζει ότι 0,3% ίσως να σχετίζεται με την αλλαγή τη δειγματοληπτική. Υπάρχει άλλος συσχετισμός που οδηγεί στην αύξηση του ποσοστού σφαλμάτων. Θα ήθελα απάντηση από το ελεκτικό συνέδριο. Στην αρχή της εκθέσεως το ελεκτικό συνέδριο αναφέρει ότι τα διαπιστωθέντα σφάλματα δεν οφείλονται σε απάτες. Στη χώρα μου, στη χώρα που εκπροσωπώ, αν δεν ακολουθείς τους κανόνες περί δημοσίων προμηθειών, αν ζητήσεις χορηγίες για μη επιλέξιμα προγράμματα και προσπαθείς να σου επιστραφούν χρήματα για μια επιλέξη με δαπάνε μπορεί αυτό να αποκληθεί απάτη και να διωχθεί. Ποιο είναι ο ορισμό που έχει για την απάτη το ελεγκτικό συνέδριο. Την τελευταία πενταετία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορούσε τα κράτη-μέλη για τα σφάλματα. Όμως υπάρχουν σημαντικά ποσοστά σφαλμάτων σε τομεί όπου υπάρχει άμεση διαχείριση πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορεί να απαντήσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να εξηγήσει γιατί υπάρχει τέτοιο ποσοστό σφαλμάτων σε αυτού του τομείς. Το ποσοστό σφαλμάτων είναι 4,8%. Το ελεκτικό συνέδριο όμως αναφέρει ότι σε κάποιους τομείς το 60% των δειγμάτων που ελήφθησαν επηρεάζονται από τα σφάλματα. Αυτό μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι μόνο 4,8% του προπολογισμού δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά. Διότι σε κάποιους κανονικούς οργανισμούς, όταν πάει σε 60% των δειγμάτων με ατασταλίες, πρέπει να επεκτείνεις το πεδίο δειγματοληψία. Δεν νομίζω ότι έχει τέτοιο χρόνο στη διάθεσή του το ελεκτικό συνέδριο. Αυτό επηρεάζει τελικά αποτελέσματα όμω και τα ποσοστά ασφαλμάτων. Την εκτίμηση των ασφαλμάτων για το σύνολο των δαπανών και για όλο τον προπολογισμό. Σχετικά με τις οικονομικές διορθώσεις. Με ανησυχία διαβάζω σελίδα 28 της εκθέσεως που αναφέρεται ότι μία διόρθωση έπρεπε να γίνει από την Ισπανία. Ανταυτού, η Ισπανία έπρεπε να υποβάλει κι άλλες εκθέσεις περί δαπανών για να μπορέσει να ζητήσει τη διόρθωση. Τι λέμε, ότι αν δεν πάρουμε τα χρήματα με τον ένα τρόπο τα παίρνουμε με άλλο. Αυτό δεν είναι οικονομική διόρθωση. Δεν εφαρμόζεται η αρχή της διόρθωσης. Το λεκτικό συνέδριο αναφέρεται στην αύξηση προχρηματοδότηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο ισολογισμός δείχνει ότι τα πως... η προχρηματοδότηση ανέρχεται στα 57 δισεκατομμύρια ευρώ, 40% του προπολογισμού δηλαδή, πολλά χρήματα, που δεν δικαιολογούνται πώς χρησιμοποιούνται. Θεωρείται ενεργητικό, αλλά δεν ξέρουμε πώς δαπανάται. Το ε, ελεκτικό συνέδριο λέει ότι αυτό το ποσό προχρηματοδότησης που αυξάνεται αυξάνει και το κίνδυνο σφαλμάτων. Τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούμε αύξηση στον προπολογισμό. Και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την ροή του ρευστού και τις πληρωμές που πρέπει να καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο είναι το θέμα. Πώς εξετάζεται η προχρηματοδότηση. Ζητά το λεκτικό συνέδριο σωστή ροή του ρευστού. Εγώ δεν νομίζω ότι αισθάνομαι άνετα να εγκρίνω να χορηγηθούν άλλα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανησυχώ για αυτό το θέμα τα τελευταία πέντε χρόνια. Τι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συνάδελφοι είπαν ότι θέλουν ένα σχέδιο δράση, ένα πρόγραμμα και ότι πρέπει να βρούμε λύση. Σχεδόν στο τέλο τη θητείας μου πρέπει να πω ότι η μόνη λύση που διαβλέπω είναι οι ευρωβουλευτέ για μια φορά να αρνηθούν να δώσουν απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή. Δηλαδή να χρησιμοποιούνται σωστά τα χρήματα των φορολογουμένων. Αυτή είναι η ευθύνη της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος και ο προτελευταίος από τις πολιτικές ομάδες είναι ο κύριος Ζέντεργαρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ το ελεκτικό συνέδριο Πολύ ενδιαφέρον το έγγραφο αυτό. Το λάβαμε μόλις χθες το απόγευμα όμως. Και είναι και αρκετά ογκώδες το έγγραφο θα έλεγα. Διαβάζοντάς το όμως, ρίχνοντας το μια ματιά, αυτό που ξανά εκπλήσει, διότι είναι σαν να τα έχουμε δει όλα και κάτι το παρελθόν, déjà vu δηλαδή, το πιο συγκλονιστικό όμως είναι η σύνοψη που υπάρχει. Εκεί που αναφέρεται στη μεικτή, στην κοινή διαχείριση οι αρχές των κρατών μελών είχαν αρκετές πληροφορίες να διορθώσουν τα σφάλματα. Και αυτό είναι μια δήλωση η οποία με συγκλονίζει. Ας αφήσουμε παράμερα για την ώρα το ότι κάποιες χώρες διαλύονται μπροστά στα μάτια μας και οι κρατικοί μηχανισμοί τους. Τα περισσότερα όμως κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να χειρίζονται τα προγράμματα και θα μπορούσαν να το κάνουν. Θα μπορούσαν να είχαν ανακαλύψει και να είχαν διορθώσει τα σφάλματα. Αυτό αναφέρεται. Δεν το έκαναν όμως. Εφόσον περί αυτού πρόκειται, πρέπει να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Γιατί έγινε αυτό. Αν πουλούσε την παλιά καλή εποχή ένα βράχο στη Δύση, στην Άγρια Δύση, αυτό θα ήταν απάτη, αναμφισβήτητα. Αλλά εδώ έχουμε παραδείγματα γεωργικής στήριξης για δασοκομεία ή για ορεινές περιοχές. Εξού και οι ερωτήσεις που προκύπτουν. Έχουμε παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία το ελεκτικό συνέδριο θεώρησε ότι ήταν αναγκαίο να κληθεί η Όλαφ, να επιληφθεί του θέματος η Όλαφ, διότι το ελεκτικό συνέδριο θεώρησε ότι δεν επρόκειται επί ανεπαρκούς εφαρμογής κανόνων ή ε, έλλειψη διοικητικών πόρων κλπ. Αλλά ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είχαν παραβιαστεί κανόνες για να αποκτηθούν επιδοτήσεις, διότι αυτό είναι απάτη. Απάτη που έχει διαπραχθεί κατά του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Άρα είναι θέμα που αφορά την Όλαφ. Καταλαβαίνω βέβαια ότι το ελεκτικό συνέδριο δεν έχει την εξουσία, δεν είναι εξοπλισμένο να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Υπάρχουν όμως τέτοια παραδείγματα. Το ελεκτικό συνέδριο κάποια δεδομένη στιγμή κάλεσε την Όλαφ διότι είχε υπόνοιες διάπραξης απάτης. Έχουμε μακροσκελή κατάλογο παραδειγμάτων που παρατίθεται. Και το ελεκτικό συνέδριο υποθέτει φαντάζομαι ότι έχουν διαπραχθεί σφάλματα καλή την πίστη. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση που ανέφερα. Έχω δεύτερη ερώτηση για το ελεκτικό συνέδριο. Κάπου αναφέρεται ότι 38% των συναλλαγών που ελέγχθησαν εμπεριέχουν σφάλματα. Μικρά σφάλματα, μεγάλα σφάλματα, σφάλματα όμως. Κάποια από τα σφάλματα θα μπορούσαν να μην επηρεάζουν τις πληρωμές κατά πολύ και τον προϋπολογισμό. Όμως το ελεκτικό συνέδριο θα ήθελα να μου πει πιστεύετε ότι το 38% είναι σωστό ποσοστό, σωστό στοιχείο ότι βασίζεται επί της μεθόδου ελέγχου. Αν εξετάσετε όμως τις ίδιες συναλλαγές, έχετε τη γενική εντύπωση εξετάζοντας συναλλαγές, γιατί αυτή είναι η δική μου εντύπωση, ότι δύο από τις πέντε συναλλαγές εμπεριέχουν σφάλματα. Έχουμε κάποια εξήγηση γι' αυτό. Διότι είναι πολύ μεγάλο ποσοστό σφαλμάτων στα δείγματα που έχετε πάρει. Ε, αυτό είναι το δεύτερο ερώτημα. Τρίτο ερώτημα που έχω. Το ελεκτικό συνέδριο έχει κάποια εξήγηση γιατί πηγαίνουμε προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, έχουμε αύξηση του ποσοστού σφαλμάτων. Γιατί. Διότι ακούω πολλά σωστά επιχειρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι άκουσα όλα τα θετικά στοιχεία και πριν και τα επιχειρήματα. Ξανά τα έχουμε δει αυτά. Ντεζά βίου και πάλι. Η μόνη εξήγηση που έχω στο μυαλό μου είναι ότι κάτι έκτακτο συνέβη. Έχουμε κάτι καινούριο που συνέβη. Έχουμε νέα επιχειρήματα. Έχετε κάτι νέο να μας πείτε που να δικαιολογεί την αρνητική τάση που διαπιστώνετε; Διότι αυτό είναι πρόβλημα. Η τάση είναι πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο φέτος, πέρσι ή πρόπερσι αυτά τα χρόνια. Πραγματικότητα είναι ότι έχουμε επιστρέψει στα επίπεδα του 2008. Έχουμε περίπου τα ίδια ποσοστά σφαλμάτων όπως με το 2008 και ήταν εποχή υλικών, ε, εκλογών. Θα το βελτιώσουμε αυτό. Ο κ. Σεμέτα το 2010, θυμάμαι, μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έλεγε ότι με τα χαρά διαπίστωνε ότι υπήρχε μια μείωση του ποσοστού σφαλμάτων. Και τότε θεωρούσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει καλή δουλειά. Όμως επιστρέψαμε πάλι στα ποσοστά του 2008 και έχουμε και άλλες εκλογές και πάλι που επικίνδυνε. Και αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Δεν είναι το έτος το συγκεκριμένο και μόνο. Ευχαριστώ τον κύριο Σέντεργατ. Και τέλος, κύριο Χάουζερ, Πάρα πολύ σύντομα θα μιλήσω κι εγώ. Τρία ερωτήματα. Στη σελίδα 11, στην σύνοψη του γερμανικού κειμένου, αναφέρονται 678 εκατομμύρια τα οποία συμπεριλήφθηκαν στις ανακτήσεις του 2012, αλλά έχουν πράγματι ανακτηθεί τα από αυτά και περιλαμβάνονται. Ε, είναι τα χρήματα αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί τα χρήματα αυτά τα οποία θα έπρεπε να είχαν πράγματι ανακτηθεί μέσα στο χρόνο αυτό. Τα 678 περιλαμβάνουν αυτό λοιπόν και το δεύτερο πόσο είναι τα κονδύλια αυτά τα οποία συνολικά πρέπει να ανακτηθούν και σε ποιους τομείς είναι τα πόσα αυτά τα οποία είναι υπό ανάκτηση. Θα ήθελα τώρα να δώσω πάλι το λόγο στον κύριο Καλντέρα και στον κύριο Σεμέτα και μετά μπορούμε να περάσουμε σε ένα δεύτερο γύρο. Έχουμε άλλους τέσσερις συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο, αλλά πρέπει βέβαια <clears throat> να έχουμε χρόνο για να προλάβουμε να, να, να κάνουμε και αυτή την, το δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Καλντέρα. Θα προσπαθήσω και εγώ όσο μπορώ να αντιμετωπίσω τα πολλαπλά αυτά ερωτήματα τα οποία έχουν διατυπωθεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για τα σχόλια και τις ερωτήσεις τους. Προσπαθήσω να ακολουθήσω τη σειρά των ερωτήσεων και σε ορισμένε περιπτώσεις θα προσπαθήσω να συνδέσω ομοειδή ερωτήματα γιατί πολλά από αυτά επαναλήφθηκαν από πολλούς ομιλητές. Ο κύριος Πίπα ζήτησε ζήτησε από το ελεκτικό συνέδριο να ε, προχωρήσει σε ελέγχους αναχώρα και να κάνει πιο λεπτομεριακή παρουσίαση στην έκθεσή του. Εγώ το έχω συζητήσει ήδη προηγουμένως με τον κύριο Πίπερ. Το πιστοποιητικό αξιοπιστίας δεν είναι σχεδιασμένο για να δίνει μία λεπτομερή έκθεση για κάθε μία από τις 27 χώρες τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, άμα είναι θέματα που αφορούν ειδικά ένα κράτο θα πρέπει να αντανακλώνται, αλλά αυτό θα γίνει από το ελεκτικό συνέδριο επί τη βάση μια κατανομής ανθρωπίνων και υλικών πόρων για, την, ε, για τις ενέργειες αυτές. Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να κατανοήσω την ε, απογοήτευσή σας για το συνοπτικό σημείωμα για το πιστοποιητικό αξιοπιστίας στο επίτομο κείμενο είναι θέμα παρουσίασης, τα ίδια πράγματα λέγονται όπως λέγονται και πέρσι, είναι συμπεπυκνωμένο κείμενο, δεν είναι πλήρης περιγραφή όπως πέρσι, ίσως είναι λιγότερο ορατά, ίσως είναι θέμα σελειδοποίησης και ίσως του χρόνου μπορούμε να το βελτιώσουμε αυτό. Κύριε Βόν, μιλήσατε για τις διορθώσεις της ε, δημοσιονομικές διορθώσεις για ορισμένες χώρες. Ε, δεν ξέρω αν και αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί από ορισμένους συναδέλφους μου. Αλλά είναι πολύ πλοκό το θέμα αυτό. Όταν προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε αυτά τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει ο πειρασμός να πει κανείς να πιστέψει ότι αυτά τα οποία αναφέρονται στην ε, έκθεση της Κομισιόν για την υποστασία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης δεν συνάδουν με τα ποσά που αναφέρει το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όμως με αυτόν τον τρόπο εποφελώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες ερμηνείες αντιμετωπίζονται τα θέματα αυτά από διαφορετικές οπτικές γωνίες που έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προστατεύσει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κάνει με αποτελεσματικό τρόπο. Το ελεκτικό συνέδριο είναι υποχρεωμένο να παρουσιάσει το επίπεδο των σφαλμάτων που βρισκούν οι λογιστικοί του έλεγχοι. Το γεγονός ότι οι περισσότερες διορθώσεις που αναφέρονται από την Κομισιόν αναφέρονται σε χρονικές εποχές που είναι από το 1994 έως το 2006, ενώ εμείς αναφερόμαστε στο 2012 στο, στην έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι συγκρίσιμα. Τότε ήταν πολύ υψηλότερα τα ποσοστά σφαλμάτων στο διάστημα 1996 μέχρι 2006. Από το 2006 και μετά μειώνονται τα ασφάλματα, τα δύο-τρία τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί λιγάκι, αλλά σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσιονομικές περιόδους τα ασφάλματα έχουν μειωθεί. Τότε, λοιπόν, το 1994 με το 2006 ήταν υψηλότερο το ποσοστό ασφαλμάτων. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε την είναι αξιόπιστη της προσπάθειας της Κομισιόν και πρέπει να την παροτρύνουμε να συνεχίσει τις προσπάθειές της. Το να έχουμε δημοσιονομικές διορθώσει. αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται τα ασφάλματα. Ήδη αναφερθήκαμε σε μια σε ορισμένε τέτοιε περιπτώσει. Αν δεν υπάρχει καθαρό αποτέλεσμα, τα σφάλματα παραμένουν. Είναι διαφορετικό το να προστατεύσουμε τον προϋπολογισμό και είναι διαφορετικό το θέμα του αν ξεπερνιούνται τα σφάλματα. Εάν λοιπόν ένα κράτος μέλος αποκομίζει κάποια ωφέλη ε, ουσιαστικά οι διορθώσεις μεταφέρουν ποσά από ένα δικαιούχο σε κάποιον άλλο. Ποιος πληρώνει σε τελική ανάλυση. Ο φορολογούμενος το κάνει, ο εθνικός φορολογούμενος. Γιατί προστατεύουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αλλά σε κάποιο βαθμό ο προπολογισμό αυτό υποστηρίζεται από του εθνικού φορολογούμενου. Μπορούμε να προστατεύσουμε λοιπόν τον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωση, αλλά αυτό δεν είναι ταυτόσιμο με την εξάλληψη των σφαλμάτων. Οι διορθώσει χρειάζονται χρόνο για να είναι αποτελεσματικέ. Μιλήσαμε για την περίπτωση της Ισπανίας. Πόσο καιρό χρειάστηκε αυτή η αλλαγή για να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι αυτές οι διορθώσεις προέρχονται από την προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο και χρειάζονται χρόνο για να υλοποιηθούν. Συνολικά θα έλεγα ότι οι δημοσιονομικές διορθώσεις μας δίνουν μονάχα ένα κομμάτι της συνολικής εικόνας. Μας καταδεικνύουν τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται από την Κομισιόν για να για να διορθωθούν τα σφάλματα που υπάρχουν και να ανοιχνευτούν τα χρεωστήτως κατά δευληθέντα. Η πλήρης εικόνα όμως εμφανίζεται μόνο στο έργο του ελεκτικού συνεδρίου που ελέγχει σε ποιο βαθμό ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα πανάτια σωστά και τι μπορούμε να πούμε για αυτό το 2012 και έρχομαι στο ερώτημα των σφάλματων. Τα σφάλματα βέβαια δεν είναι σφάλματα λόγω απάτης. Δεν ταυτίζονται αυτά. Και ο έλεγχος μας δεν έχει σαν στόχο να ανακαλύψει απάτες. Η απάτη είναι μία ηθελημένη πράξη για να αποκομίσει κανείς κάποιο όφελος, ενώ ένα σφάλμα δεν είναι πάντα ενσυνείδητο. Αν βρούμε όμως μια περίπτωση όπου υπάρχει υποψία απάτης, προφανώς θα παραπερθεί στο αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν δοθεί λοιπόν τέτοια στοιχεία στην Όλαφ, η οποία όλα βέβαια μετά πρέπει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Αλλά μια ατασταλία <clears throat> σημαίνει ότι δοθήκανε κάποια χρήματα χωρίς να έχουν ακολουθηθεί πλήρως οι κείμενοι κανόνες. Αλλά αυτό δεν ισοδυναμεί πάντα με μία απάτη. Όταν λοιπόν ε, έχουν, δεν έχουν ακολουθηθεί πλήρως οι κανόνες. Τώρα, <coughs> τώρα το τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε πιο μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τις ταμιακές ροές. Το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι η Κομισιόν έχει ήδη τις απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με τις συνάψεις υποχρεώσεων, τις πληρωμές, την προχρηματοδότηση, όλα αυτά τα στοιχεία που επιτρέφουν στην Κομισιόν να προχωρήσουν σε λογικό επίπεδο και να έχουν κάποιες προβλέψεις για τις μελλοντικέ ανάγκες πληρωμών. Όλα αυτά καταγράφονται ήδη στους ισολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να προβλέψει τις απαιτούμενες ταμιακές ροές. Βέβαια υπάρχουν τα λεγόμενα RAL, τα ρεσταλικίδε, τα υπολοιπόμενα ποσά. Και η Κομισιόν το απεικονίζει αυτό πολύ σαφώς στις εκθέσεις Κάθε χρόνο τα ποσά αυτά τα οποία παραμένουν εκκρεμή αυξάνονται. Αν δείτε το κενό του 2007-2013 βλέπουμε ότι το αρχικό χάσμα των 50 δισεκατομμυρίων έχει διπλασιαστεί σχεδόν. Είμαστε στα 114 δισεκατομμύρια. Το ποσό αυτό λοιπόν που έχει να κάνει με την προετοιμασία για πληρωμές δεν ήταν επαρκές για να μειώσει το χάσμα αυτό. Και αυτό φυσικά οδηγεί σε μεγαλύτερα ερωτήματα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Εγώ κατανοώ αυτά τα οποία αναφερθήκατε στα οποία αναφερθήκατε για το Ευρωελεκτικό Συνέδριο. Σήμερα συζητάμε για την ε, ετήσια έκθεση βέβαια μονάχα, αλλά λαμβάνω υπόψη όλες τις παρατηρήσεις σας. Τώρα, για τις ε, <clears throat> αυξήσεις στα ποσοστά ασφαλμάτων. Τονίστηκε ότι υπήρξαν αυξήσεις και στον τομέα του πρώτου πυλώνα στη Γεωργία. Εδώ νομίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Κομισιόν για να εντοπίσουν τις ρίζες του προβλήματος αυτού. Το ελεκτικό συνέδριο θεωρεί ότι υπήρχαν οι συνθήκες οι οποίες θα οδηγούσαν σε ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων. Για κάποιο λόγο δεν έχει γίνει αυτό πραγματικότητα. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι δεν λειτουργεί σωστά. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν υπάρχει σύστημα λειτουργικό εντοπισμού των προβλημάτων στα κρατη σε ορισμένα κράτη-μέλη, αυτό είναι ένα πρόβλημα και η Κομισιόν πρέπει να επιληφθεί του θέματος αυτού και αυτό ίσως να δικαιολογεί κάποια από την αύξηση στο ποσοστό σφαλμάτων συμφωνήσαμε ότι δεν πρέπει σήμερα να αποδηθούμε σε μια συζήτηση επί της μεθοδολογίας. Δεν έχει αλλάξει η μεθοδολογία του ελεκτικού συνεδρίου, απλώς έχει ενημερωθεί και επικαιροποιηθεί ακολουθώντας τις ε, τροποποιήσεις στο σύστημα α, ε, λογιστικού χαρακτήρα που λειτουργεί βάσει δεδουλευμένο και απεικονίζει την πραγματικότητα, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Έχουμε τώρα μια ενημέρωση του συστήματος που μπορεί να εξασφαλίσει μια συγκρισιμότητα σε όλους τους τομείς πολιτικής και να έχουμε και μεγαλύτερη συγκρισιμότητα όπως έχετε ζητήσει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. <clears throat> Δεν αλλάζουμε λοιπόν κάθε χρόνο τη μεθοδολογία μας, ούτε κάθε δύο χρόνια, ούτε κάθε τρία χρόνια. Το ελεκτικό συνέδριο είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για τους λογιστικούς ελέγχους, παραμένουμε ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος λειτουργεί με επαγγελματικό τρόπο, αν αλλάξουν τα διεθνή πρότυπα ή χρειάζονται βελτίωση και εμείς θα πρέπει να τα παρακολουθήσουμε στον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τους δικούς μας λογιστικούς ελέγχους. Οποιαδήποτε τροποποίηση σε ό,τι αφορά το πιστοποιητικό αξιοπιστίας θα πρέπει να τύχει συζήτηση μαζί σας με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο. Όλα αυτά λοιπόν δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι αποτελούν ευνηδιαστικές ενέργειες. Το ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε για τις ε, ανακρίβειες για τα ποσοστά σφαλμάτων απαιτεί, ένα, μια, απαιτεί μια απάντηση και πρέπει να το πω σαφώς, δεν πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα του ελεκτικού συνεδρίου δεν αποκλίνουν από αυτά που ζητά ο δημοσιονομικός κανονισμός και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Και εσείς παίξατε ένα ενεργό ρόλο στη δημιουργία του νέου δημοσιονομικού κανονισμού. Προβλέπει μια διαδικασία κατά μεταξύ των ελεκτών και του ελεκτικού συνεδρίου. Με αυτή τη διαδικασία μπορεί να υπάρξει η ευκαιρία για τους ελεκτές να δώσουν νέα στοιχεία. Και είναι καθήκον του ελεκτικού συνεδρίου όταν έρθουν τα νέα αυτά στοιχεία, <clears throat> τα οποία έχουν έγκυρο χαρακτήρα, έχει καθήκον το ηλεκτρικό συνέδριο να λάβει υπόψη τα νέα αυτά στοιχεία. Και αυτό έχει συμβεί σε ορισμένε περιπτώσει, όταν οι εθνικέ αρχέ ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνουν πρόσθετα στοιχεία κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας κατά αντιπαράθεση πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και πιστεύω ότι ότι οι περιπτώσεις αυτές οι οποίες θεωρούνται ότι μπορεί να περιέχουν κάποιο σφάλμα ή κάποια ατασταλία δεν, <clears throat> που δεν θεωρήθηκε ότι ήταν σημαντικές, αν έρθουν νέα στοιχεία λαμβάνονται και αυτές τις περιπτώσεις υπόψη στον υπολογισμό για το ποσοστό σφαλμάτων. Και όλα αυτά με την διαδικασία αυτή συνεννόησης. Πρέπει λοιπόν στο έργο μας να λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά τα πρόσθετα στοιχεία που μας δίνουν οι Εθνικές Αρχές και η Κομισιόν και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο πηγάζει από τα επαγγελματικά μας πρότυπα. Τελευταίο σχόλιο σε σχέση με το ερώτημα της κυρίας Αντριάσεν. Αν η αύξηση των σφαλμάτων οφείλεται στην αλλαγή της ε, διαδικασίας στιγματοληψίας. <clears throat> Νομίζω ότι μόνο ένα μικρό τμήμα μπορεί να οφείλεται σε μια αλλαγή της ε, διαδικασίας δειγματοληψίας και το είπα και στην αρχή. Και φυσικά υπάρχει το δειγματοληπτικό σφάλμα πάντα. Αν θέλετε να συγκρίνετε λοιπόν το 2011 με το 2012 με επί της ίδιας βάσης η αλλαγή είναι μονάχα από το 3,9 στο 4,5 και όχι στο 4,8. Κύριε Ζόντεργατ, όταν αναφέρεστε στην συχνότητα των σφαλμάτων και την εκτίμηση των σφαλμάτων, του ποσοστού σφαλμάτων, στο δικό μας δείγμα, που είναι περιορισμένο βέβαια, το ποσοστό σφαλμάτων, το ποσοστό των περιπτώσεων που βρήκε μία ατασταλία το συνέδριο. Δεν κάνουμε προεκβολή. Κάνουμε προεκβολές μονάχα όταν έχουμε σοβαρά σφάλματα και από αυτά προσπαθούμε να δούμε τι συμβολή θα είχαν στο ποσοστό σφαλμάτων. Η συχνότητα λοιπόν των σφαλμάτων είναι σημαντική για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ποιοι είναι οι τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερος ελοχεύων κίνδυνος. <clears throat> Και πράγματι είναι συνήθως περιοχές που έχουν να κάνουν με την πολιτική συνοχής και την αγροτική ανάπτυξη σε ό,τι αφορά τις περιοχές κοινή διαχείρισης με τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω τώρα αν έχω ξεχάσει κάποια ερωτήματα. Είμαι έτοιμος να σας δώσω στη συνέχεια γραπτές απαντήσεις αλλά προς το παρόν κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Μόλις μίλησα με τον Επίτροπο τον κ. Σαμέτα, μπορεί να μείνει λίγο περισσότερο. Uh, Έχουμε άλλους τέσσερις επίγνωτες στο λόγο, οι οποίοι προτείνουν να λάβουν από ένα λεπτό το λόγο, ώστε να Να δούμε τι έχει να, πει, τι ο κύριος Καλτέρα. Κυρία Αγιάλα πρώτη. Πρόεδρε, κάπως μας απογοητεύει το ότι μας δώσετε μόνο ένα λεπτό, γιατί ναι, θα ήθελα να πω κάτι για τον κύριο Πίπερ, για μια που δεν συμφωνώ με κάποια από αυτά τα οποία μας εξήγησε. Αυτά τα οποία είπε είπε κάτι, μετά ξεκαθάρισε κάποια άλλα θέματα του κ. Καλτέρα και είπε μετά ότι είχαμε κάποιε αλλαγέ στη δημοτοληψία που έχουν να κάνουν με κάποιε αλλαγέ, κυρίω όσον αφορά τι εξωτερικέ σχέσει κλπ. Και μα είπε ο κ. Καλτέρα ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια γενική άποψη του τοπίου, αλλιώ η απλούστηση που κάνουμε δεν θα είναι ρεαλιστική. Έχουμε κάποιε λεπτομέρειε εδώ που είναι σημαντικέ. Έχουμε α πούμε κάποια παραδείγματα που αφορούν το κοινωνικό ταμείο, τελείως συμπτωματικά, ε, αφορούν την Ισπανία και για 3 έως πέντε χρόνια πήγαν αυτά. Έρχεται η Τρόικα όμως, μας ζητάει εργασιακή μεταρρύθμιση και ε, λέμε για απολύσει ενώ είπαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν συμβάσει εργασία ενό έτου. Το 2008 ξεκίνησε η κρίση. Να, επομένω ότι εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα έλλειψης ευελιξίας. Κύριε Σεμετά, λάβετε το αυτό υπόψη. Τι γίνεται με τους κανονισμούς με το 2007, του Φεντέρ και των άλλων υπήρξε κάποια προσαρμογή στην κρίση, αλλά αυτό το οποίο θέλαμε ήταν τα επιδόματα ενεργείας να φτάσουν τα 5 χρόνια, αλλά στην ε, Ισπανία πού να βρει κανείς δουλειά. Ε, ούτε για ώρες δεν βρισκούμε εύκολα. Επομένως, όσον αφορά τώρα τι γίνεται με τους συνήθεις υπόπτους που είπε ο κύριος Πίπερ για την Ισπανία και την Ελλάδα και τους συνήθεις υπόπτους γενικώ. Για κοιτάξτε τι έγινε στο 2012. Θυμάμαι ότι όσον αφορά την προστασία του προπολογισμού και όσον αφορά κάποιες ε, αναστολές και κάποιες ε, διακοπές το 2012 εμείς διεκπαιρεώσαμε κάποιες περιπτώσεις τέτοιες. Καταφέραμε να έχουμε κάποιες επιδόσει καλύτερες από τη Γερμανία. Γιατί η Γερμανία τότε είχε πολύ περισσότερες αναστολές και διακοπές. Άρα, κύριε Πίπερ, να δούμε όλο το τοπίο και ο καθένας τέλο πάντων ασχολείται περισσότερο μετά του οίκου του. Κάτι άλλο τώρα. Όταν λέμε για τα επιμέρου ποσά, του επιμέρου τομείς του προπολογισμού και λέμε για Ισπανία, για Ελλάδα, για σχέ... χώρες συνοχής και βλέπουμε ότι όλοι αυτοί προσφεύγουν στο ΦΕΝΤΕΡ. Πώς γίνεται όμως αυτό. Όταν έχουμε μια χώρα που παίρνει 50 και κάνει 5 λάθη είναι 10%. Μια χώρα που παίρνει 5 και κάνει λάθος 3, τότε έχει λάθος 33%. Οπότε βλέπετε ότι πολλές φορές αντιστρέφουμε τις συνέπειες του ποσοστού λάθους. Άρα όλα είναι θέμα του πώς θα παρουσιάζει κανείς πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Τρία λεπτά μιλήσατε εσείς. Καλώς πάντων. Επόμενος ο κύριος ε, Κάλφιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Άρα εγώ πλην δύο λεπτά. Και έτσι θα εξισορροπήσω. Θα προσπαθήσω να είμαι πραγματικά σύντομος. Βεβαίω και έπρεπε να λάβουμε κάποια μέτρα μετά την ανάλυση της έκθεσης και ευχαριστώ την ε, κύριο Καλντέρα. Πριν φτάσουμε πάντως σε κάποιο είδους συμπεράσματα θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι γίνεται με τα λίγη της μεθοδολογίας. Οι αλλαγές δεν, δεν, δεν είναι αλλαγές κάθε αυτές, είναι το ότι αλλάζουμε πολύ συχνά πράγματα και αυτό το οποίο εγώ δεν έχω πάρα πολύ καλά είναι τι γίνεται με τις προκαταβολές, τι γίνεται με τις εξωτερικές δράσεις, τι γίνεται με την έρευνα, πώς είναι η μεθοδολογία επιδράει από αυτόν, γιατί κατά τα άλλα αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίζεται σε κάθε βασικό πρόγραμμα της Ένωσης. Επίσης, είπατε ότι έλαβαν ε, υπόψη ε, ότι είναι ποσοτικά αποτιμήσιμα τα λάθη των ελευθερισμών οργανών. Όμως, για πέστε μας, ακριβώς ποιες είναι οι επιπτώσεις για κάθε τομέα τον οποίο εσείς ε, τον ελέγχετε. Γιατί έχουμε, έχουμε δυσκολίες να προσαρμοστούμε στην κάθε φορά νέα μεθοδολογία. Δεύτερον, προτείνατε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτούς τους πίνακες σε σχέση με προηγούμενες επιδόσεις και προηγούμενες συστάσεις. Διαπιστώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν ληφθεί μέτρα κατόπιν των ε, ε, συστάσεών σας και ακόμα υπάρχει πρόβλημα που μας θα πρέπει να κάτσουμε για να αναλύσουμε <coughs> τι γίνεται άπαξ και έχουμε τις ε, συστάσεις και την υλοποίησή τους γιατί τα πράγματα είναι έτσι. Και αυτό το οποίο δεν έχω καταλάβει αυτό που είπατε πρόεδρε είπατε για 270 δις που είναι πιστός υποχρεώσεων και είπατε ότι αυτά δεν εκταμιέστηκαν, δεν απορροφήθηκαν. Τέλο πάντων δεν κατάλαβα τι έγινε εκεί. Επίσης για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο έχουμε αυτήν την προσέγγιση με βάση τις δαπάνες, έχουμε τώρα τις συμφωνίες εταιρικών σχέσεων κλπ. κλπ. Εν ώψη 2020 πολύ σημαντικό. Όταν λέτε για το 4,8 πόσο στο λάθος. Τι πάει να πει. Αφορά το σύνολο του 140 δις τότε πάμε 6,7 δις που πλήσονται από τα λάθη. Τι είναι, υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ε, επιπτώσεων. Τέλο πάντων τα λάθη επιδρούν σε δύο επίπεδα του συνόλου. Κάτι άλλο τώρα εδώ που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το κοινοβούλιο. Αν μπορείτε, συγκρίνετε με το προηγούμενο πλαίσιο. Νομίζω ότι ο τρόπος που γίνονται οι δαπάνες εξηγεί τις διαφορές. Πάμε το 7,3 και πάμε στο 3,3 το 2009. Τα λάθη και τώρα έχουμε ξανά αύξηση. Για να κάτσουμε να συγκρίνουμε με το προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο για να δούμε πώς, πώς μας συγκρίνουμε το, το, το, την ίδια τακτική και διαφορετικά αποτελέσματα. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λουκίου Σέπιν, θα προσπαθήσω να σπάσω το ρεκόρ των προλαλήσάντων. Να είμαι συντομότερος. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω απευθυνόμαι στον κύριο Μούλτερ ότι το 2004, Οκτώβριο του 2004 ήταν το τελευταίο θετικό δελτίο αξιοπιστία όταν ανέλαβε Επίτροπο Και ήμουν στο γραφείο του επιτρόπου που πρέπει να το εφαρμόσει αυτό και θυμάμαι το 2006 το επίπεδο σφαλμάτων ήταν 7,5% το ποσοστό. Εγώ θεωρώ ότι στη φύση του προπολογισμού έγκυται το πρόβλημα. Έγινε προσπάθεια μέσω μικροδιαχείρισης στην Ευρώπη να επιτευχθεί ε, σωστή διαχείριση. Και σε κάποιους τομείς που ήταν προβληματικοί όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος, Έχουμε επιδοτήσεις εκεί σε αυτούς τους τομείς, έχουμε σειρά προγραμμάτων, στόχων, έχουμε το πρόγραμμα SMART, 52 στόχοι περιέχονται και μόνο 8 είναι προσμετρήσιμοι. Αυτό δεν είναι κάτι που οδηγεί σε καλή κατάτηση προπολογισμού, αυξάνει το ποσοστό σφαλμάτων, υπάρχει συσχετισμός μεταξύ κακής εφαρμογής μέτρων και κακής δίκησης και συμφωνώ με την ιδέα του εισηγητού, δηλαδή να υπάρχει ένα σύστημα κυρώσεων που θα επιβάλλεται. Πρέπει να δούμε όμως και πού φταίμε και εμείς. Κάποια μέλη της Επιτροπής αυτής είναι και μέλη της Επιτροπής Προπολογισμών και βλέπουμε ότι στην Επιτροπή Προπολογισμών υπάρχει πίεση για περισσότερη ανάληψη υποχρεώσεων και μεγαλύτερο προπολογισμό. Άρα κάνουμε, δίνουμε περισσότερε υποσχέσει. Και όταν έχουμε έναν προπολογισμό υποσχέσεων, δεν αποτελεί έκπληξη ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Διότι έχουμε έναν προπολογισμό που συνεχώ ε, δέχεται πιέσει για τι πληρωμέ. Υποστηρίζω λοιπόν την απόφαση που ελήφθη από το Συμβούλιο. Και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων είχαν δίκιο. Χρειαζόμαστε μικρότερο προπολογισμό που θα εφαρμόζεται καλύτερα από τον παρόντα. Ευχαριστώ τέλο το ελεκτικό συνέδριο, έξοχη δουλειά που έκανε. Έγινε ένα έλεγχο τη πραγματικότητα, χρειαζόταν κάτι τέτοιο και καλωσορίζω την ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Ελπίζω ότι θα βελτιωθούν οι εργασίε. Υπ' αυτέ τι περιστάσεις όμως δεν μπορούμε να δώσουμε απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. αγαπητοί συνάδελφοι, σα ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω ότι ο πρόεδρος ε, Καλτέρα πρέπει να φύγει στις 11. Ίσως μπορεί να δώσει μια σύντομη απάντηση λοιπόν για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Και εγώ σας ζητώ συγγνώμη που θα πρέπει, θα πρέπει να φύγω. Μπορώ να σας στείλω γραπτές απαντήσεις αν θέλετε και μπορούν να εξάλλου και οι συνάδελφοί μου εδώ από το ελεγκτικό συνέδριο ίσως να αναφερθούν στα θέματα αυτά. Ε, εάν το επιθυμείτε, μονάχα ένα σύντομο σχόλιο για την ε, σύγκριση με προηγούμενες δημοσιονομικές ε, περιόδους. Για μένα το πιο σημαντικό, πιο σημαντικό μήνυμα που προσπαθώ να σας ε, μεταφέρω φέτος με την ετήσια μας έκθεση είναι ότι δεν πρέπει να κοιτάμε προς τα πίσω, αλλά να κοιτάμε προς τα μπρος. Έχουμε μια νέα προγραμματική περίοδο που έρχεται, υπάρχουν νέοι κανόνες οι οποίοι έρχονται σε εφαρμογή νέες προτεραιότητες, νέα σχέδια. Πρέπει να έχουμε απλά συστήματα, σαφείς στόχους, ε, δείκτες απόδοσης οι οποίοι μπορούν να δώσουν κάποιο απτό αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι το εγχείρημα το οποίο θα κάνει καλύτερο το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δόντως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλύτερες ευκαιρίες να παρακολουθήσει όλα αυτά τα στοιχεία και νομίζω ότι <clears throat> με αυτή την ιδέα στο μυαλό σας θα πρέπει να αξιολογήσετε τις προσπάθειές μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν και συγγνώμη που πρέπει να φύγω. Okay, thank you very much, President Caldera. Σας ευχαριστούμε Πρόεδρε Καλδέρα. Uh, συνάδελφοι, ο συνάδελφος Σάββα ήθελε να πάρει το λόγο. Είναι ο τελευταίος συνάδελφος που έχει τη δυνατότητα για να δώσουμε μετά το λόγο στον Επίτροπο ούτως ώστε να απαντήσει στα όσα υπόθηκαν. Πάνω από 12 συνάδελφοι μίλησαν. Ο κύριος Σαβαρή λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Λυπόμαι που καθυστέρησα, είχα σημαντική έκθεση στην Επιτροπή Μεταφορών κ. Καλτέρα απεχώρησε. Ευχαριστώ όμως το Ελεκτικό Συνέδριο για τη δουλειά που έκανε. Να σας πω τι γίνεται με τους διάφορους οργανισμούς, γιατί λάβαμε τις περισσότερες αιτήσεις έκθεσης. Ένα-δύο πράγματα μου προσήλξαν την προσοχή. Πρώτα απ' όλα, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα καινοτομία και Τεχνολογίας εξέδωσε μια αιτιολογημένη άποψη το Ελεκτικό Συνέδριο για την ανεπαρκή ποιότητα των πιστοποιητικών ελέγχου. Αυτό αφορά τις δαπάνες για διάφορες χορηγίες. Μετά το Frontex. Ανεπαρκή στοιχεία για τον έλεγχο περί ατασταλιών κλπ. Και για τις διάφορες συναλλαγές που αφορούσαν τις χορηγίες στον τομέα. Άλλο ένα θέμα. και έχουμε νέο οργανισμό. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για Υποστήριξη Ασύλου με το δίκτυο οργανισμών υπήρχε έξοχη συνεργασία. Και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει η εργασία μας κάπως να συντονιστεί. Το καλοκαίρι αποφασίσαμε ότι όλοι οι αποκεντρωμένοι φορείς θα ετοιμάζουν και θα υποβάλουν εκθέσεις τακτικά και οι προθεσμίες. Προσπαθούμε να κάνουμε πιο ευκάμπτες διαδικασίες. Και θα πρέπει να υπάρχει προθεσμία υποβολή ερωτήσεων για τις ε, τους οργανισμούς για τις απαλλαγές, 26 Νοεμβρίου. Μετά έχουμε τους Κιώδης. Θα τα καταφέρουμε αρχές Νοεμβρίου, την πρώτη εβδομάδα ε, αρχές Δεκεμβρίου, συγγνώμη, 2 με 5 Δεκεμβρίου να το καταφέρουμε αυτό. Και μετά πάμε προς ακροάσεις. Θα διεξαχθούν είτε στις 20-21 Ιανουαρίου. Αναφέρω τις ημερομηνίες. Τέλος λέει ο κ. Σαβραμά. Υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που μπορούμε να κατονομάσουμε που θα προσκληθούν στην ακρόαση. Το δίκτυο, ο συντονιστής του δικτύου, η ERA, μετά οργανισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων και δύο οργανισμοί που προανέφερα που είναι κάτω από το μεγεθυντικό φακό η ΕΤΑΡΗ και το Frontex και μετά το, το Frontex και μετά ο Οργανισμός στην υποστήριξη του ασύλου. Πρέπει να μάθουν και αυτή τη διαδικασία και οι νέοι φορείς. Και οργανισμοί που κατά το παρελθόν ανεβλήθη ή απερίφθη απαλλαγή πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. Τι διορθώσεις έχουν κάνει. Η ΣΥΠΟΛ, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία Ασφαλείας Τροφίμων, η ΕΦΣΑ και ο Οργανισμός Φαρμάκων. Και αυτούς θα θέλαμε να τους καλέσουμε σαν Και η CDC ενδεχομένως. υπήρξε γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου. Κατά την άποψή του είχε επιληθεί το πρόβλημα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτος να αναφερθεί στον οδικό χάρτη. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Τι θα εξετάσουμε όσον αφορά τις απαλλαγές των διαφόρων οργανισμών. Ευχαριστώ και πάλι το ελεγκτικό συνέδριο για την δουλειά που έκανε στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι είχαμε μια πλούσια συζήτηση, αναφέρθηκαν πολλά σημαντικά στοιχεία και τα οποία απαντήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Φυσικά πολλά από αυτά συνάπτονται και με την Κομισιόν και θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Σεμέτα να παρουσιάσει τη δική του θέση ως εκπροσώπη της Κομισιόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για τις ερωτήσεις τους. Θα ήθελα να ξεκινήσω με γενικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου του ελεκτικού συνεδρίου, πάνω από 130 δις ευρώ δαπανήθηκαν σωστά. Σημαντικότατο. Πρέπει να υπογραμμιστεί. Να ληφθεί υπόψη. Δεύτερον, δεν έχουμε συγκρίσεις με κράτη-μέλη. αν τα πηγαίνουμε καλύτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, φάση δαπάνη του προπολογισμού από τα κράτη-μέλη. Δεν έχουμε συγκρίσιμα προγράμματα στα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχουν κράτη-μέλη που εφαρμόζουν την ίδια μεθοδολογία από το λεκτικό συνέδριο και αξιολογούν ότι ο τρόπο τι εθνικέ δαπάνε με παρόμοιου κανόνε. Αν γινόταν αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε συγκρίσει. Αλλά δεν γίνεται. Και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αν τα πάει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα δαπάνε. Σε πρόσφατη διάσκεψη εκπρόσωποι των ΗΠΑ είπαν ότι το ποσοστό σφαλμάτων του είναι παρόμοιο με το δικό μα. Κάτι άλλο σημαντικό. Το υπογραμμίζω. Δεν μιλάμε για τα λογιστικά και τους λογαριασμούς δεν υπάρχουν σφάλματα στα λογιστικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έκτο, έβδομο χρόνο, έκτο χρόνο κατά σειρά. Και σε οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία, αν είναι ξεκάθαρα το λογιστικά, δίνονται σαφείς πληροφορίες επενδυτές για τη θέση της εταιρείας. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι λοιπόν όσον αφορά τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και δεν είναι εύκολο να γίνουν οι λογαριασμοί διότι και τα λογιστικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι είναι πάρα πολύ ε, πολλά τα χειρήματα πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του υλοποίησης του προπολογισμού. Αυτά που είπε ο κ. Πίπερ τώρα. Συμφωνώ πλήρως με την προσέγγισή σας όσον αφορά τους τέσσερις στόχους που θέλετε να θέσετε στη διαδικασία της απαλλαγής. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας. Επί όλων αυτών, όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της πρώτερης απαλλαγής. Υπάρχουν διάφορες συστάσεις που εφαρμόστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρθρο 318 και σχετική έκθεση που υποβλήθηκε πολύ πιο έγκαιρα από ό,τι άλλες χρονιές και όσον αφορά και το περιεχόμενο των εκθέσεων που πρέπει να βελτιωθεί και βελτιώθηκε σημαντικά. Δεν θα σταματήσουμε όμως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα μάλιστα επεξεργάζεται ένα πλήρες σύστημα αναλύσεως επιδόσεων. Εκεί θα συμπεριλαμβάνεται η πλήρης αλυσίδα. Από τα σχέδια μέχρι τις εκθέσεις δραστηριοτήτων, συνοπτικές εκθέσεις και αξιολόγηση και έκθεση αξιολόγησης. Και έτσι θα εξετάζονται όλα αυτά και θα συντονίζονται. Συμφωνώ με τα σχόλιά σας. Πρέπει πράγματι να έχουμε τη σωστή δομή όσον αφορά τη μέτρηση των επιδόσεων. Χρειαζόμαστε προσέγγιση που να σχετίζεται άμεσα με τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Σημαντικότατο. Πρόθεσή μας είναι να το κάνουμε αυτό ακριβώς. Πολλές ερωτήσεις αφορούσαν τις οικονομικές διορθώσεις, αν ελήφθησαν δεόντως υπόψη ή όχι και τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Πρώτον, που θέλω να τονίσω, το παρόν σύστημα οικονομικών διορθώσεων εφαρμόζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο δεν μπορούμε να εφεύρουμε κάτι που δεν ταιριάζει με την νομοθεσία. Και η ισχύουσα νομοθεσία ακριβώς τονίζει ότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει οικονομική διόρθωση και συμφωνεί ένα κράτος μέλος με τη διόρθωση αυτή, τότε μπορεί να ξαναχρησιμοποιήσει τους πόρους για άλλα προγράμματα. Διότι προβλέπεται αυτό στην νομοθεσία. Αυτό το σύστημα έχουμε επί του παρόντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προστατεύουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, επιβάλλοντας οικονομικές διορθώσεις. Διότι αυτές οι δαπάνες των κρατών μελών που δεν είναι σωστές ή εμπεριέχουν σφάλματα πρέπει να διορθωθούν. Επιβάλλεται. Το επιβάλλουμε αυτό. Και αυτά τα προγράμματα αποκλείονται από χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό προπολογισμό. Η κυρία Γκρέσλε είπε ότι δεν συμφωνεί με το ότι προστατεύουμε τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά δεν προστατεύουμε τους εθνικούς προπολογισμούς μέσω, οικονομικών διορθώσεων. Πρέπει όμως να δώσουμε ευθύνες και στα κράτη-μέλη μας και στα κοινοβούλια αυτών. Και αυτά πρέπει να λάβουν υπόψη ότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε οικονομική διόρθωση στο κράτος μέλος και το κράτος μέλος δεν ανέκτησε τα χρήματα από τους τελικούς δικαιούχους, τότε πιθανότατα το Εθνικό Κοινοβούλιο πρέπει να εξετάσει την κατάσταση. Και να το αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σχετικά με το μέλλον Γνωρίζω πολύ καλά ότι η μελλοντική νομοθεσία για την επόμενη προγραμματική περίοδο προβλέπει καθαρή οικονομική διόρθωση. Και η παρούσα νομοθεσία προβλέπει αυτού του είδους τη διόρθωση σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις όπου το κράτος μέλος διαφωνεί με την οικονομική διόρθωση. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει αυτή την οικονομική διόρθωση. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις συμφωνούν τα κράτη-μέλη με τις οικονομικές διορθώσεις. Στην επόμενη προγραμματική περίοδο, εάν εγκριθούν οι κανόνες όπως προβλέπετε, αυτή θα είναι πολύ αυστηρότερη Σύμφωνα με αυτούς, όταν μετά την υποβολή των λογαριασμών ανακαλυφθεί ότι υπάρχουν ατασταλίες όσον αφορά τις δαπάνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να επιβάλλει οικονομική διόρθωση. Άκουσα πολύ προσεκτικά τα σχόλια του κυρίου Πίπα, του εισηγητού, για την ανάγκη αυτοματισμού όσον αφορά αυτή η δικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό επεξεργάζεται. Ένα σχέδιο κατά εξουσιοδότηση πράξης ετοιμάζει στα πλαίσια της μελλοντικής νομοθεσίας. Θα έχουμε έτσι δυνατότητα να καλύψουμε τις ιδέες που εκφράσατε κύριε Σιγητά στην ε, παρέμβασή σας. Όσον αφορά τους κακούς μαθητές όπως αποκαλούνται και αρκετά κράτη-μέλη που αποτελούν την πλειοψηφία όσον αφορά τα σφάλματα, δημιουργούν τα περισσότερα σφάλματα, ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε σχέδια δράσης για αυτές τις χώρες, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Κατά χώρα. Γεωργία παραδείγματος χάρη. Ο συνάδελφός μου, ο Επίτροπος ο Τσόλας, συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη όσον αφορά συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση αδυναμιών που εντοπίστηκαν τα τελευταία χρόνια, μάλλον στην περασμένη έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Εμείς ως πολιτικοί βέβαια θέλουμε άμεσα αποτελέσματα από τη δράση. Πρέπει όμως και να είμαστε ρεαλιστές. Οι δράσεις που δρομολογούνται από τα κράτη-μέλη χρειάζονται χρόνο. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και θα δώσουν αποτελέσματα μετά από κάποια χρονική περίοδο, όχι αμέσως. Πιστεύω όμως ότι δράσεις που εφαρμόζονται τώρα είναι καθοδόν θα συμβάλλουν στη μείωση του ποσοστού σφαλμάτων στο μέλλον. Ηρίστον παρόδο, άμα μιλάμε για την Ισπανία, συγκεκριμένα οι Ισπανικές αρχές επί τη βάση των σχεδίων δράσεως Ήδη άλλαξαν κάποια επιχειρησιακά προγράμματα όσον αφορά τον περίπλοκο χαρακτήρα των κανόνων επιλεξιμότητας. Και αυτό αντιστοιχεί και στην υπερβολική νομοθεσία που ανέφερε ο κύριος Γκάιερ στην περσινή έκθεση. Και αυτά τα θέματα ήδη εξετάζονται ήδη από τις εθνικές αρχές, συγκεκριμένη περίπτωση από τις ισπανικές αρχές. Και αυτό νομίζω ότι απαντά και στο ερώτημα της κυρίας Αγιάλα Σέντερ όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα που έφυξε για δαπάνες των κοινωνικών ταμείων και όρους για την χρήση αυτών. Αυτοί ήταν εθνικοί οι κανόνες. Δεν ήταν κανόνες που επευλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν κανόνες που επέβαλαν οι εθνικές αρχές και δεν σεβάστηκαν τους κανόνες αυτούς και αυτό αποτελεί και μία έκκληση προς τα κράτη-μέλη να απλουστεύσουν τους κανόνες για την απασχόληση. Και όπως είπα στην εισαγωγή, τα κράτη-μέλη εκείνα που χρησιμοποιούν τις νέες δυνατότητές μας με απλουστευμένα μοντέλα όσον αφορά το κόστος αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο σφαλμάτων από τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν το περίπλοκο σύστημα και τους σχετικούς κανόνες. Ο κ. Στάς ζήτησε να ετοιμάσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των αδυναμιών. Αυτό μπορούμε να το επεξεργαστούμε. Να δούμε τα βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν περαιτέρω για να βελτιωθεί η κατάσταση. Μετά, όσον αφορά την αλλαγή μεθοδολογίας, Δεν αμφισβητούμε τις μεθοδολογικές αλλαγές του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι δική του ευθύνη. Όμως, οι αλλαγές αυτές επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα, τα γενικά αποτελέσματα, τα συνολικά, κυρίως όσον αφορά την άμεση διαχείριση, όπου εφαρμόστηκαν οι νέοι κανόνες. Παραδείγματος χάρη, αν το λεκτικό συνέδριο ακολουθούσε ίδια προσέγγιση. Όπως παλιά, στις εξωτερικές σχέσεις ή την έρευνα, τότε και στους δύο τομείς η κατάσταση θα ήταν βελτιωμένη εν συγκρίση με τα προηγούμενα χρόνια και το συνολικό ποσοστό ασφαλμάτων και στις εξωτερικές σχέσεις και στην έρευνα θα ήταν κάτω από το υλικό όριο τους, που έχει θέσει το ελεκτικό συνέδριο. Ε, οι εξωτερικές σχέσεις από το 3,3% σφάλματος το 3,2% από αυτό οφείλεται στις αλλαγές της μεθοδολογίας. Στην έρευνα από το 3,9% γενικό ποσοστό σφάλματος το 2,2% προέρχεται από την αλλαγή μεθοδολογίας. Άρα είναι σημαντικός αντίκτυπος στον τομέα της άμεσης διαχείρισης. Οι μεθοδολογικές αλλαγές έλαβαν χώρα κυρίως εκεί. Να πω και κάποια ακόμα. Ο Γιάνν Μιλντερ αναφέρθηκε στον τομέα της γεωργίας και μας είπε ότι αυξάνεται το ποσοστό των λαθών για τη Γεωργία και επίσης ε, είπαμε ότι μας προβληματίζει επίσης αυτό το θέμα και είπαμε ότι οι συνάδελφοι συνεργάστηκαν εντατικότατα με τα κατημέρια για να μπορέσουν να δουν τι γίνεται ε, με αυτά τα προβλήματα. Οπότε όταν έρθει η ώρα της ακροασίας του θα σας εξηγήσει κατά λεπτό την κατάσταση. και όσον αφορά αυτά τα καινούργια μέσα και να δούμε τα κάτι όσον αφορά αυτήν την ε, το, αυτή την πολιτική, την πολιτική γεωργίας που είναι ακριβώς ε, περισσότερες δαπάνες μας τώρα. Για να δούμε κάτι που είπε η κυρία Άντρεσεν για τα αμέσα σφάλματα, τη διαχείριση. Έχει γίνει εδώ πέρα όντως μια τέτοια αύξηση και αυτό βασικά αφορά την αλλαγή της μεθοδολογίας ε, χωρίς αυτήν την ε, αλλαγή είπαμε ότι θα είναι τα πράγματα πολύ θα ήταν τα λάθη πολύ λιγότερα και επίσης να μην ξεχάσουμε αυτά που είπε το ηλεκτροσυνέδριο συνέδριο όσον αφορά την προχρηματοδότηση για τις εξωτερικές σχέσεις. Εν προκειμένου θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι οι εξωτερικές σχέσεις είναι ο μόνος τομέας όπου οι συνομοθέτες συνεφώνησαν να υπάρχει η δυνατότητα της προχρηματοδότησης χωρίς να υπάρχει κάποιο είδου εκαθάριση ενδιάμεση. Και αυτό εν μέρη εξηγεί γιατί έχει αυξηθεί η προχρηματοδότηση για αυτά τα θέματα. Ε, επίσης, πάνω κάτω τα είπαμε όλα. Α, για, ε, για την απαλλαγή είπε και ο κύριος Βόνος, αναφορά τη μέτρηση των επιδόσεων. Νομίζω σας εκάλυψα και σύντομα θα διαπιστώσετε ότι έχουμε αυτό το, το έγγραφο το οποίο εντέλει τις υπηρεσίες για το τι θα κάνω όσον αφορά την αλυσίδα διαχείρισης και ελέγχου της Επιτροπής. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπελίου Πρόεδρος για αυτές τις κατελητικές σας παρατηρήσεις. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Πίπερ, ο συγητής μας. Πάρα πολύ σύντομα λέει ο κύριος Πίπερ. Όλα αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι νομίζω ότι δείχνουν την ε, γενική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ μας. Φυσικά θα πρέπει να συζητήσουμε πιο λεπτομερώς και να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις σε ορισμένα σημεία. Εγώ δεν θέλω τώρα να ε, να καταφερθώ κατά της Ελλάδος ή της Ισπανίας αλλά αναφέρω, αναφέρθηκα σε ένα αυτοματισμό ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει όλες τις χώρες. Και η Γερμανία, η ε, Βόρεια Ιρνανία, Βεσφαλία και η Ζαρλάνδη και αυτές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν με αυτόν τον τρόπο, με αυτοματισμό, εάν υπήρχαν, εφόσον υπάρχουν τόσο πολλά σφάλματα. Μιλήσα λοιπόν για ένα αυτοματισμό και όχι για καταγγελία μονάχα ορισμένων χωρών. Για ε, την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου ε, είπε ο κ. Καλτέιρα ότι δεν δέχεται να υπάρξουν εκθέσεις σε επίπεδο χωρών αλλά υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν και μια ομοσπονδιακή δομή όπως είναι η Γερμανία και οι χώρες αυτές όπως είναι η Γερμανία, όπως η Ισπανία που έχουν αυτόνομες κυβερνήσεις και ομοσπονδιακή δομή θα ήταν χρήσιμο να εξεταστούν λίγο καλύτερα. Θα μας έδινε αυτό πολύ περισσότερα στοιχεία. Θέλω επίσης να επιβεβαιώσω αυτά που λέει ο κύριος Επίτροπος. Το 95% είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε θετικά. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να δώσω κι εγώ. Αλλά για το 5% που παραμένει όπως και στο 75-80% ήταν πάντα οι ίδιες χώρες που είχαν τα περισσότερα σφάλματα. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ακόμα και αυτό το τελευταίο 5% παρά το γεγονός ότι είναι μόνο 5% και να μην το ξεχάσουμε. Και πάλι λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω όλους που ε, συμμετέσχαν σε αυτή τη συζήτηση, να ευχαριστήσω και το Ελεκτικό Συνέδριο και την Κομισιόν. Σίγουρα θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία απαλλαγή. εφέτος. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος, τον εισηγητή. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο τέλο τη ε, συνεδρίασής μα σήμερα το πρωί και ευχαριστώ όλους οι οποίοι ήταν παρόντες. Ευχαριστώ και τον πρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου και τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου και τον κύριο Σεμέτα. Φυσικά θα ακολουθήσει η διαδικασία απαλλαγής που θα μας οδηγήσει να εξετάσουμε πιο προσεκτικά πολλά με μονομενα στοιχεία. Μας ενδιαφέρει όλους να μειώσουμε το ποσοστό των σφαλμάτων και να δούμε κατά πόσο οφείλονται όλα αυτά στην πολυπλοκότητα των κανόνων. Ίσως οι κανόνες αυτοί μπορούν να απλοποιηθούν περισσότερο. Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο έχω διατυπώσει και υποστηρίζω εδώ και πολύ χρονικό, πολλά χρόνια. Και η κυρία Γκρέσλε η οποία είναι αρμόδια για τα θέματα του προπολογισμού με τον κύριο Μπελίνη και αυτοί έχουν ζητήσει επιμόνωση να υπάρξει μια απλοποίηση στου κανόνε του προπολογισμού. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή και όλου του συναδέλφου και κλείνω το κομμάτι της, επίσης, της ανοιχτής συνεδρίασης. Ζητώ όμως από τους συντονιστές, εάν θέλουν, να παραμείνουν για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αμέσω με τη συνεδρίαση των συντονιστών. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ όλους τους καλεσμένους να αποχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ.